Okay, please take your seats. Παρακαλώ καθίστε. Sorry to be delayed. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Because I was simply waiting for uh, the coordinators. Περίμενα να μαζευτούν οι συντονιστές. Thank you. Can I point out that the... Ευχαριστώ. Τα πρακτικά τη συνεδρίαση των συντονιστών ε, θα διανεμηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα το απόγευμα και αν δεν κάνω λάθο, αύριο είναι η έγκριση. Αύριο μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση. Ε, ρίξτε μια ματιά και μια και συζητάμε ε, κάποια θέματα τα οποία ε, καλό είναι να τα έχουμε εγκρίνει πριν εγκρίνουμε τα πρακτικά. Πέστε μας οτιδήποτε υπάρχει. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 για την κατάσταση των θαλασσών. Έχουμε τη δεύτερη έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση θα συζητήσουμε τι Μεσόγειο και τον έξινο Πόντο. και θα ήθελα και ζήτησα μάλλον και μια έκθεση προέδρου για την διακήρυξη της Μάλτας ε, Medfish Forever. Έχουμε τη Βάλερη Λέιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε όλοι στη Μεσέγειο και τον Εύξηνο Πόρντου, το Mare Θα ξεκινήσω από μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα της Μεσογείου είναι γνωστό πως ε, υπάρχουν αρκετές ε, ιδιαιτερότητες ε, στη λεκάνη της Μεσογείου. Το γεγονός ότι σε βιολογικούς όρους υπάρχει μεγάλη βιοπικιλότητα, πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες λεκάνες. Υπάρχει επίσης και ένα πολύπλοκο θαλάσσιο οικοσύστημα και υπάρχουν και κάποια είδη τα οποία ενδημούν μόνο στην ε, Μεσόγειο. Έχουμε ε, πάνω από 2.500 αποθέματα, μια ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει για παράδειγμα στον Ατλαντικό. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει όπως ε, στον Ατλαντικό για παράδειγμα αποκλειστική οικονομική ζένη, κάποιες κοινοτικέ ζώνες όπως τις αποκαλούμε στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχουν πολλά κοινά αποθέματα επίσης, πολύ μεγάλος αριθμός αποθεμάτων και κάποια δεν ανήκουν μόνο στα κοινοτικά ύδατα, αλλά και σε άλλες τρίτες χώρες της Μεσογείου. Επίση, υπάρχει και μια διεθνή συνιστόσα. Η πλειοψηφία αυτών των ε, ε ε, αποθεμάτων ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης της Επιτροπής ε, Διαχείρισης των Βαθύβιων Ιδών της, της Μεσογείου. Έχουμε 26 χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη σύνθεση του στόλου. Στο Μεσόγειο υπάρχει μια μεγάλη σύνθεση στόλου και ένα μεγάλο σκέλος αποτελείται από μικρά σκάφη τα οποία φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν ε, στους λιμένες, εκφορτώνουν μικρές ποσότητες αλευμάτων και επομένως υπάρχει και η διαφορά εδώ σε σχέση με τον Ανατλαντικό όπου είναι πιο βιομηχανικός ο στόλος ε, και οι εκφορτώσεις είναι σε πολύ σημαντικούς όγκους. Ε, επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες οι οποίες σχετίζονται και με κάποια πολιτική αστάθεια που υπάρχει στη Μεσόγειο. Ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετές ε, σειράξει ε, στη Λιβύη, στη Συρία. Ε, υπάρχει όμως και στο Εύξηνο Πόντο το θέμα της Κρυμαία και της Ρωσίας. Υπάρχει και ένα πρόβλημα που αφορά και στον ε, περιορισμό των θαλάσσιων ζωνών και επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας, αλίας αγιουγιού, γιατί πολλά ε, πράγματα γινόντουσαν χωρίς κανέναν έλεγχο σε διεθνή ήθατα στο παρελθόν. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί όταν πρέπει να διαχειριστούμε τα αποθέματα της Μεσογείου πρέπει να λάβουμε όλες αυτές τις διατηρότητες υπόψη. Πρέπει να τα έχουμε κατά νου και σε επίπεδο διαχείρισης αλλά και σε επίπεδο των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της αλίας. Δυστυχώ, έχουμε διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια ότι μειώνονται οι θαλάσσιοι πόροι της Μεσογείου και η μείωση οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, ε, κυρίως ε, στην υπεραλίευση, ε, τις δραστηριότητες ε, λαθρέας άναρχης και παράνομης αλίας, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εναρμονισμένα σχέδια διαχείρισης των αποθεμάτων, κυρίως για τα κοινά αποθέματα. Υπάρχει επίσης πολλαπλασιασμός των δραστηριοτήτων, ε, κυρίως ε, σε ε, ναυτιλία, τουρισμός, εκμετάλλευση φυσικού αερίου, ρήπανση, ρήπανση πλαστικών που είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, και υπάρχει και η χορύπανση. Θα επανέλθω και σε αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει αντίκτυπο και αυτό στα αποθέματα. Και ε, όλα αυτά, όπως σας είπα, σημαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω και της υπεραλίευσης. Τώρα, όσον αφορά τον εύξηνο πόντο, Υπάρχουν εκεί κάποιες ιδιαιτερότητες που αφορούν και πάλι τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μια θάλασσα που είναι ημίκλειστη όπως και η Μεσόγειος. Ε, και υπάρχει και το εξής. Δεν υπάρχει οξυγόνο όπως υπάρχει σε άλλες λεκάνες. Δηλαδή, το 90% των υδάτων της ε, Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ 100 και 200 μέτρων, είναι ανοξικά, δηλαδή δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν οξυγονώνεται η θάλασσα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και ασθενή βιοποικιλότητα, ελάχιστα αποθέματα, 8 αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εμπορία ε, στον εύξηνο ε, πόντο, το καλκάνι, ε, καρχαρίες ε, σκουμπρί, μπαρμπούνια και τρία-τέσσερα άλλα. υπάρχει πρόβλημα επίσης λαθρέας αναρχής και ανα... παράνομης αλληλείας. Ε, όπως σας είπα υπάρχουν και γεωπολιτικά βρήματα τα οποία ε, παρακολύουν τη διαχείριση των θαλασσιών πόρων και υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την κλιματική αλλαγή. Επομένως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη λεκάνη, τα χαρακτηριστικά και πάλι είναι ε, το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντική η παραλίευση και εδώ δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα. Ε, υπάρχει ε, καταμερισμός των υδάτων για όλα την ε, περιοχή του Ευξηλουπόντου. Τώρα, Κατάσταση των αποθεμάτων. Η κατάσταση των αποθεμάτων, όπως γνωρίζετε, είναι σε μια κατάσταση λόγω της υπεραλίευσης. Ε, η πλειονότητα των αποθεμάτων ε, της Μεσογείου και του Ευξήνου Πόντου υπεραλιεύονται. Κατά μέσο όρο έχουμε 2,2 FMSY για το σύνολο των αποθεμάτων. Ελάχιστα ε, αποθέματα είναι στο MSY, στα Αναταλικά έχουμε μπαρμπούνι και γάβρο και στην ε, Εύξηνο Πόντο έχουμε δύο είδη τα οποία βρίσκονται σε MSY, αλλά η σαρδελόραγκα, η παπαλίνα και ένα ακόμα είδος ε, και ε, από εκεί και πέρα Όσον αφορά ε, τα επιστημονικά στοιχεία, η πλειονότητα των στόλων ε, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά τις δυνατότητες αλίευσης που έχουν. Και όπως ε, βλέπετε και στη διαφάνεια υπάρχει πάρα πολύ σημαντική υπεραλίευση. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ε, κάπως θετικές. Αν δείτε το τέλος της καμπύλης υπάρχει μια αύξηση της βιομάζας ε, και επομένω. Ε, ε, το ΣΑΚ που είναι το επιστημονικό ε, όργανο της CGPM το διαπιστώνει αυτό και επομένως παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα βρίσκονται σε ικτρή κατάσταση έχουμε ένα κάπως πιο αισιόδοξο μήνυμα και οι επιστημονικές ενδείξεις μας δείχνουν ότι είναι διατηρήσιμη υπερεκμετάλλευση. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουμε υπερελίευση, ε, διατηρούνται τα αποθέματα χωρίς ε, να ε, μειώνονται δραματικά. Πρόκειται και αυτό για μία ιδιαιτερότητα της Μεσογείου, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις αποθεμάτων που είναι σαφείς και το αποδεικνύουν και τα στοιχεία. Γιατί αν δείτε τα στοιχεία του CGPM, CGPM Είχαμε το 2003 2 εκατομμύρια τόνους εκφόρτωσης. Σήμερα στο 2016 μάλλον έχουμε 1,3 εκατομμύρια τόνους. Έχουμε λοιπόν μείωση των εκφορτώσεων. Διαπιστώνουμε επίσης ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό απορρίψεων. Οι απορρίψεις είναι πάνω από 275.000 τόνους στη Μεσόγειο και επίσης ε, αυξάνονται οι ε, τα ποσοστά κάποιων ειδών που είναι ευαίσθητα. Όσον αφορά τα αλλιεύματα, τα μικρά πελαγικά είδη έχουν τους πιο σημαντικούς όγκους στη Μεσόγειο. Και όσον αφορά τα αλλιεύματα, το δυτικό σκέλος είναι το πιο παραγωγικό. Έχουμε 272.000 τόνους εκφόρτωσης και μετά έχουμε την Αδριατική θάλασσα. Τώρα, όσον αφορά στόλους και εκφορτώσεις, ο πιο σημαντικός στόλος είναι ο τουρκικός, ο ιταλικός, ο στόλος της Αργερίας, της Ελλάδος, της Τινησίας και της Κροατίας, για να έχετε μία εικόνα για την αναλογία κατανομής των ε, αλλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο. Τώρα, όσον αφορά τι κοινωνικο-οικονομικέ πτυχέ που είναι πάρα πολύ σημαντικέ, παρά το γεγονό ότι υπάρχει υπεραλίευση, παρά το γεγονό ότι ε, κάποια πράγματα είναι λιγότερο σημαντικά, ε, είναι σημαντικά τα ποσά της αλληλεία. Στη Μεσόγειο έχουμε ε, πάνω από 86.000 ε, σκάφη και κυρίως ε, τέσσερις χώρες έχουν 17% η Τουρκία, 17% η Ελλάδα, 15% η Τινησία και 13% η Ιταλία. Ε, η μικρή κλίμακα αλίας φυσικά είναι πολύ σημαντική. 70.000 σκάφη στη Μεσόγειο που είναι το 50% των εσόδων και το 60% της απασχόλησης και έχουμε 2,8 δις δολάρια κύκλο εργασιών και η απασχόληση είναι 240.000 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, η Ευρώπη όσον αφορά το στόλο της έχει 50% του ευρωπαϊκού στόλου που αλλιεύει στη Μεσόγειο, που είναι περίπου το 38% της ε, ευρωπαϊκής υποσχόλησης και 12% των εκφορτώσεων. Τα έσοδα είναι σχετικά σταθερά για τους ε, Ε, παραγωγούς. Κροατία, Μάλτα και Κύπρος είχαν μια μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ε, παρά το γεγονός ότι είναι χαμηλό το ποσοστό των εκφορτώσεων, ε, φαίνεται να υπάρχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο λόγω της αυξημένης τιμής των αλλιευμάτων ε, στη Μεσόγειο σε σχέση με άλλες λεκάνες. Και επίσης ε, το επιχειρησιακό κόστος είναι πολύ μικρότερο στη Μεσόγειο από ό,τι σε άλλες λεκάνες και αυτό γιατί είναι παράκτια η αλία και επομένω χρησιμοποιούν λιγότερη, λιγότερα καύσιμα για την αλία. Όταν λοιπόν ένα αλληλεία ε, έχει τρία κασόνια ψάρια, έχει βιώσιμη αλληλεία ε, στη Μεσόγειο, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει στην, ε, στον Ατλαντικό. Επομένως διατηρείται η οικονομική δραστηριότητα και στο παρελθόν αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι δεν χρειάστηκε να υποχρεώσουμε το στόλο αυτό να κάνει αναδιόρθρωση και να λάβει μέτρα. Πιστεύω όμως ότι αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Το γεγονός ότι στη Μεσόγειο δεν υπήρχαν ε, σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, ότι ο στόλος μπορούσε να επιβιώσει, διότι πρόκειται για μικρούς στόλους και όπως σας είπα τα εισοδήματα ήταν εξορροπημένα, ε, σημαίνει ότι η νομοθεσία και οι επιστημονικές νομοδοτήσεις ε, επικεντρώθηκαν περισσότερο στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Που τι σημαίνει αυτό, ότι όσον αφορά την νομοθεσία, διαπιστώνει κανεί ότι στην ιστορία τη νομοθεσία, είτε πρόκειται για κοινοτική είτε για διεθνή νομοθεσία, υπήρχε ελάχιστη νομοθεσία. Ο πρώτο κανονισμό για τη Μεσόγειο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε το 1994 και έλαβε υπόψη του μόνο κάποιε διατάξει ε, για το άνοιγμα των δικτυών, την προστασία των οικοτόπων ε, και το ελάχιστο μέγεθος για την εμπορία. Μετά υπήρξε ένας δεύτερος κανονισμός το 2006, ο οποίος καθόριζε και ένα καθεστώς ε, ε, αλλιευτικών πόρων, αλλά πάντα αποκεντρωμένο και το διαχειριζόντουσαν τα κράτη-μέλη και δεν υπήρχε λοιπόν ε, νομοθεσία πέραν αυτών των καθαρά τεχνικών κανονισμών που αφορούσαν μόνο ε, κάποιες ιδιαιτερότητες της και όχι την αλία αυτή καθευτή. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην Γενική Διεύθυνση δεν υπάρχει τμήμα για τη Μεσόγειο. Το πρώτο τμήμα για τη Μεσόγειο εμφανίστηκε το 2008, δεν υπήρχε πριν. Που σημαίνει ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμίσουμε και να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα πέραν αυτών που υπήρχαν σε τοπικό επίπεδο, ε, διότι προφανώ και υπήρχαν τοπικά μέτρα. Τα κράτη-μέλη είχαν εγκρίνει κάποια μέτρα σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία υπήρχαν κάποια ε, μέτρα από τον αρμόδιο οργανισμό, που ε, τον Πριντομή, ο οποίος ε, ε, είναι πάρα πολύ τοπικός και επίσης στην Ισπανία υπήρχαν κάποιες συνομοσπονδίες, συνεταιρισμοί που διαχειριζόντουσαν την αλία. Επομένως δεν φαινόταν να υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστούν τα αποθέματα. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των μέτρων που υπήρχαν δεν έφταναν για να ρυθμιστεί η υπεραλίευση. Και όπως σας είπα, διαπιστώσαμε σιγά σιγά ότι άρχισαν να μειώνονται οι πόροι και χρειάστηκε κάπως καθυστερημένα αλλά έγινε, το Φεβρουάριο του 2016 ε, θεωρήθηκε ότι απέτυχαν όλα αυτά τα μέτρα και ο κύριος Βέλα έκανε ένα σεμινάριο στην Κατάνια που είχε συμμετοχή όλων των επιστομιών αρμόδιων για τη Μεσόγειο και αρχέ των κρατών μελών για να διαπιστωθεί η επιτυχία των μέτρων που είχαν ληφθεί και ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την υπεραλίευση και την επίτευξη του μέγιστου βιώσιμου αποθέματο του MSY. Ο κύριο Βέλα λοιπόν τότε λόγω αυτή τη αποτυχία αποφάσισε να συγκαλέσει υπουργική διάσκεψη τον Απρίλιο του 2016 με όλε τι χώρε τη Μεσογείου Στι Βρυξέλλε, λοιπόν έγινε μια μεγάλη σύνοδος με όλες τις χώρες τη Μεσογείου, οι οποίες ε, παραδέχτηκαν και αυτές ότι έχει από τύχη και η ε, λεκάνη της Μεσογείου αλλά και ο Ευξηνός Πόντος. Ε, ελήφθη λοιπόν η απόφαση να αλλάξει η κατάσταση, να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και συνεργάστηκαν για να εγκρίνουν τη λεγόμενη ε, δήλωση Medfish Forever το 2017 και επίσης για τον Ευξηνό Πόντο υπάρχει η διακήρυξη της Σόφιας. Τι είναι αυτές οι διακήρυξεις. Θα πείτε ότι είναι απλές δηλώσεις. Αυτή τη φορά όμως αποφασίστηκε να υλοποιηθούν μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων αυτό το οποίο αποφασίστηκε λοιπόν από όλου του υπουργού είναι ένα επίσημο μέτρο να υπάρχει μια νέα διακυβέρνηση της Αλίας στη Μεσόγειο και βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες δράσεις, τέσσερις βασικές δράσεις. Ο πρώτος άξονας είναι η βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και η συλλογή δεδομένων που αποτελεί βάση για να καθορίζονται συνέχεια μέτρα διαχείρισης να υπάρχουν επίσης ε, ε, δυνατότητες διαχείρισης αλίας με μια οικοσυστημική προσέγγιση, όχι μόνο λοιπόν όσον αφορά τα αποθέματα, αλλά όσον αφορά το συνολικό οικοσύστημα και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια νοοτροπία ελέγχων και καταπολέμησης της παράνομης αλίας, καθώς επίσης και να υπάρχει με βιώσιμο τρόπο ανάπτυξη τη μικρή κλίμακα αλληλεία και τη υδατοκαλλιέργεια. Επίση, να ενισχύσουμε το πλαίσιο συνεργασία ε, μεταξύ ε, της τη νότια και τη βόρεια ακτή, καθώ επίση και τη ανατολική ακτή και να προτείνουμε ε, να εγκρίνονται μέτρα για τη διαχείριση των αποθεμάτων που είναι σε κίνδυνο, τα κάποια υποθέματα τα οποία θεωρούνται και συμβολικά και σε επίπεδο της ε, περιφερειακής οργάνωσης, της EGPM, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών μάλλον όλων των κρατών της Μεσογείου. Αυτά ε, μεταφράστηκαν σε κάποια μέσα της Ένωσης. Το βασικό μέσο βέβαια είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική. Εφαρμόστηκε λοιπόν η κοινή αλληλευτική πολιτική και στη Μεσόγειο και αυτό μεταφράζεται αφενός από την έγκριση του πολιετού σχεδίου με τεχνικά μέτρα, ε, καθώς επίσης και ευρωπαϊκά κονδύλια ένας πρώτος κανονισμός για τις αλληλευτικές ε, δυνατότητες, εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, αλλά επίσης και συνέχεια της εφαρμογής ε, του κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα, προστασία των οικοτόπων και επίσης υπάρχουν και κάποια ενισχυμένα προγράμματα επιθεωρήσεων, τα λεγόμενα ESCIP, τα οποία ε, διαχειρίζεται ο οργανισμό ε, του Βίγκο και αποφασίστηκε για όλη τη Μεσόγειο να υπάρχει ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων για να συντονιστούν τα μέσα ελέγχων των κρατών μελών στι διάφορε λεκάνε. Ε, πρόκειται για καινοτομία, πρόκειται για ενοποίηση των ελέγχων και των μέσων που ε, υλοποιούνται ακριβώ για να ενισχύσουν την εφαρμογή μέτρων διατήρηση που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένα συντονισμό, παρά μόνο για τον ερυθρό τόνο προφανώ που υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, αλλά δεν υπήρχε τέτοιο συντονισμό πουθενά αλλού. Έγινε επίσης μια ενίσχυση του συντονισμού με το Συμβούλιο ε, και τα περιφερειακά συμβούλια, ε, το ΓΙΝΤΑΚ και το ΜΠΙΣΑΚ, που είναι ε, τα περιφερειακά συμβούλια που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση των αποθεμάτων, γιατί το ΜΕΝΤΑΚ και το ΒΙΣΑΚ το διαβουλευόμαστε για το σύνολο των μέτρων διατήρησης και τα εφαρμόζουμε μέσω αυτών. Και επίσης ζητήθηκαν και μία σειρά από μελέτες ε, με σημαντικό προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή λοιπόν ε, ζήτησε κάποιες μελέτες ε, για να δούμε την κατάσταση των αποθεμάτων. Υπάρχει μια μελέτη για να δούμε το σύνολο των αποθεμάτων. Επίσης υπάρχουν κάποια προγράμματα, τρία προγράμματα για ανάπτυξη ζωνών προστασίας Πρόκειται για το SafeNet, το MEDA και το MANTIS, ε, τα οποία καλύπτουν ε, το σύνολο των υδάτων ε, από Ανατολή προς τη Δύση ή από τη Δύση προς την Ανατολή, αν το προτιμάτε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον προστατευμένο, την δυνατότητα των προστατευμένων θαλάσσιων ζωνών, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς από πλευρά μας αποφασίσαμε επίσης να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, καταρτήσουν εθνικά σχέδια διαχείρισης. Ε, έχουμε λοιπόν αντίστοιχα εθνικά σχέδια. Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια υπάρχουν και στρατηγικοί για την υδατοκαλλιέργεια. Τέσσερις άξονες για να δούμε τα διοικητικά θέματα, να μειώσουμε το διοικητικό άκθος και το διοικητικό φόρτο, ε, να δούμε επίσης την ε, διατήρηση των υδάτων και την υγεία των ζώων και κάποια μέτρα εφαρμογή για τις ε, δραστηριότητες και κάποιες προδιαγραφές για την εφαρμογή μιας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, εγκρίθηκε ο πρώτος χάρτη αυτής της ιστορίας όλης, ο οποίο καταρτίστηκε βάσει μιας μελέτης επιπτώσεων που ξεκίνησε το 2015, δηλαδή χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να εγκριθεί αυτό το MAP. Είναι το πρώτο σχέδιο στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την κυρία Αγγιλέρα, την εισηγήτρια, που ήταν από τους βασικούς μοχλού για την έγκριση αυτού του MAP. Και εδώ έχουμε ένα καθεστώς ε, αλλιευτικών ε, ταμείων, μείωση της αλλιευτικής προσπάθειας κατά 40% μέχρι το 2025, προκειμένου να ε, καταφέρουμε τα εμβληματικά είδη, τα πιο σημαντικά εμπορικά είδη του δυτικού σκέλους της Μεσογείου, να ε, τύχουν βιώσιμης διαχείρισης. Αυτά τα μέτρα θα μεταφραστούν σε ημέρες αλλιευσής. Έχουμε επίσης ε, ε, και κάποια επιπλέον μέτρα. Έχουμε κάποιες κλειστές ζώνες για να προστατευθούν οι γόνοι, καθώς επίσης ε, και κάποια μέτρα για την ερασιτεχνική αλληλεία και μέτρα για να στηρίζουμε τον στόλο με μόνιμες δομές και προσωρινό κλείσιμο δραστηριότητας ε, και θα υπάρχουν και κάποια τεχνικά μέτρα τα οποία θα προσαρμοστούν στην περιοχή και υπάρχουν και κάποια πολύ σημαντικά μέτρα ελέγχου, το επαναλαμβάνω αυτό, για παράδειγμα η καταγραφή των ημερών αλληλείας καθώς επίσης ε, και ε, κλείσιμο της αλληλείας όταν επιτυγχάνεται η ποσόστοση. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το νέο καθεστώς ε, για, την, ε, για τα ελευτικά ε, μέτρα θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την υπεραλίευση και να έχουμε διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται ένα τέτοιο μέσο και θεωρούμε ότι είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. Ο κανονισμός εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου του 2019, τέθησε ισχύ από τον Αύγουστο και επομένως η αλληλευτική ε, προσπάθεια και οι ποσοστώσεις θα συζητηθούν στα πλαίσια του κανονισμού για τις αλληλευτικές ε, δυνατότητες, ο οποίος θα συζητηθεί το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο των Υπουργών. Ο κανονισμό αυτό ε, για τι ελευτικέ δυνατότητε, περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα. Είναι η πρώτη φορά επίση που θα υπάρξει ένα κανονισμό για τι ελευτικέ δυνατότητε. Ο κανονισμό αυτό έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι καθορίζονται ποσοστώσεις για την ελευτική προσπάθεια και επίσης ε, ε, μέτρα διαχείρισης τα οποία ενέκρινε ο CGPM. Μέτρα για κλείσιμο για τρει μήνες, κάποια κατεπήγοντα μέτρα για τα μικρά πελαγικά τραγικά είδη για 100.000 τόνους, ποσοστώσεις για το καλκάνι, οι οποίες είναι ακόμα σε υποδιαπραγμάτευση και κάποια άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να εγκριθούν ε, λόγω των συμπερασμάτων της CGPM. Τα μέτρα αυτά συνολικά μας επιτρέπουν να έχουμε μία εφαρμογή των μέτρων σε κοινοτικό και σε τοπικό επίπεδο, αλλά επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία είναι σε διεθνές επίπεδο. Όπως βλέπετε εδώ στο χάρτη, τα περισσότερα αποθέματα είναι ε, κοινά. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της αυτά τα αποθέματα, πρέπει να βασιστεί και στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του ε, GPM και επίσης να, ε, να συντονιστεί με τους υπολείπους για να λαμβάνεται ε, απόφαση για τη διαχείριση από το σύνολο των ενδιαφερομένων. Επομένως, ε, τα αποθέματα είναι κοινά, επομένως οι λύσεις και τα μέτρα πρέπει επίσης να είναι επιμερισμένα. Γι' αυτό ακριβώς και σε επίπεδο GPM Green με κάποια μέτρα. Εδώ περνάω στο επόμενο στάδιο που είναι η υλοποίηση των μέτρων διατήρησης. Από τότε που εγκρίθηκε ε, το, ο κανονισμός είχαμε 25 συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές αφορούν ε, κυρίως ε, μέτρα διατήρησης αλλά και μέτρα ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, πούμε ότι έγιναν πολύ σημαντικές προσπάθειες για να εγκριθούμε μέτρα και σχέδια διαχείρισης. Τα σχέδια διαχείρισης αφορούν και τα πιο σημαντικά είδη στη Μεσόγειο, το καλκάνι, έχετε γαρίδες βαθέων υδάτων, παπαλίνα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια είδη τα οποία θα ε, έχουν σχέδιο διαχείρισης. Υπάρχουν κάποια μέτρα για τη στρατηγική κατά της παρανομής λαθρείας και άλλη αρχής ε, πάνω από 100.000 επιθεωρήσεις έγιναν ε, από την έγκριση του Medfish Forever ε, και ε, συνελέγησαν κάποια στοιχεία και υπάρχει παρακολούθηση από εκεί και πέρα από τα κράτη σημαία. Υπάρχει και μια στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια που είναι πάρα πολύ σημαντική στη Μεσόγειο. Επομένω, θα πρέπει να φροντίσουμε να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο και να υπάρχει και συμμόρφωση προς περιβαλλοντικούς ε, κανόνες. Υπάρχει επίσης πάρα πολύ σημαντικός ρόλος για τη μικρή κλίμακα αλίας, επομένως υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για τη μικρή κλίμακα αλία και ε, στην πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν και μέτρα τα οποία ε, συζητούνται για την, ε, το αλευτικό ταμείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τη μικρή κλίμακα αλίας, να υποστηρίξουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις, την έρευνα, την κατάρτιση, ε, την ένταξη των νέων γενεών στην αλληλεία, την αξιοποίηση των προϊόντων, τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα που έχει μικρή κλίμακα αλίας να αυτοδιαχειρίζεται ε, η μέθοδη εργασίας, ε, ο ρόλος των γυναικών, κάτι το οποίο επισημάναμε επίσης αυτή τη στρατηγική και φυσικά ο αντίκτυπος της μικρής κλίμακας αλίας στο κλίμα και στο περιβάλλον που ε, είναι κάτι στο οποίο μπορεί να συμβάλλει μικρή κλίμακα αλληλεία ε, και για τη συλλαγή δεδομένων, αλλά και γνωρίζοντα και το περιβάλλον, ε, μπορούμε να έχουμε κάποιου δείκτε για τι συνέπειε τη κλιματική αλλαγή. Όπω σα είπα, εφαρμόζονται όλα αυτά τα μέτρα. Ε, εφαρμόστηκαν επίση και κάποια μέτρα όσον αφορά τι υποστημονικέ ενδείξει. Υπάρχουν επίση και μία από τι πιο σημαντικέ επικρίσει που είχαμε στη Μεσόγειο ήταν το γεγονό ότι δεν υπήρχε συντονισμό για την έρευνα, για τα επιστημονικά στοιχεία. Και Επομένως, ε, στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας ε, ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των ερευνητικών ε, μέσων για να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε την έρευνα, να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση των αποθεμάτων και καλύτερη εικόνα για την ε, διαχείριση. Το Φόρουμ για την Επιστήμη είχε συμμετοχή πάνω από 400 επιστημόνων και αρκετές χώρες συζητήθηκαν πολλά θέματα. Το, η κατάσταση των αποθεμάτων, η έννοια του κλίματος, η έννοια της ρήπανσης, κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και ε, προχωρήσαμε πάρα πολύ στη Μεσόγειο σε θέματα συλλογής δεδομένων και νομίζω ότι αυτό ε, θα είναι κάτι θετικό γιατί θα βοηθήσει να βελτιωθεί η διαχείριση των αποθεμάτων και υπάρχει και πάρα πολύ σημαντικός ρόλος όπως σας είπα ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ο κινητήριος μουχλός σε όλες αυτές τις προτάσεις. Γίνεται συντονισμός όλων αυτών των προτάσεων βάσει των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνουμε από την Επιστημονική Επιτροπή και ε, γίνεται συντονισμός με τις χώρες ε, της Νότιας Μεσογείου αλλά και τις χώρες της, ε, του Ευξήνου Πόντου. Υπάρχουν πάρα πολλές διμερείς σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας. Η συνεργασία λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο κυρίως για θέματα παράνομης λαθρέας και ανεργής αλληλείας. Ο οργανισμός έκανε πάνω από 130 σεμινάρια κατάρτισης ε, και χάρη σε αυτές τις ε, στρατηγικές ε, προσελήφθησαν οι επιθεωρητές, υπήρξε κατάρτιση και βλέπετε ότι υπάρχει ε, δραστηριοποίηση σε όλη τη λεκάνη τη Μεσογείου. Υπάρχουν πολλέ χώρε που έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, πρέπει να αλλάξει ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στη Μεσόγειο και πώ διαχειριζόμαστε τα αποθέματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι είναι όλο και πιο παρόντε στο διεθνέ προσκήνιο για να μπορέσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμμετέχει με 4 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των GFCM, τον οργανισμό, ε, για να ε, υλοποιηθούν τα διάφορα μέτρα για τη μικρή κλίμακα για τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή και τη δειγματολοψία στη θάλασσα, γιατί αυτό είναι κάτι δαπανηρό και πρέπει κάπως να χρηματοδοτείται, αλλά επίσης για να βελτιώσουμε την έρευνα υπάρχουν ε, κάποια μέτρα για συγκεκριμένα είδη, αλλά και για τον αντίκτυπο στο κλίμα Υπάρχει επίσης ε, χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε ε, τις χώρες ε, για να μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες ελέγχους τους. Επίσης υπάρχει χρηματοδότηση σε προγράμματα ΦΑΟ, ΙΣΜΕΔ κλπ. Κάποια άλλα για να μπορέσουν αυτές οι χώρες να συλλέγουν δεδομένα, να κάνουν ανταλλαγές απόψεων όσο αφορά τα επιστημονικά στοιχεία. Επομένως, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός και αναγνωρίζεται από αυτές τις χώρες και τώρα πολύ γρήγορα να περάσω στο μέλλον. Έγινε μία διάσκεψη τον Ιούνιο, υπουργική, στο Μαρακές και στη διάρκεια αυτής της διάσκεψης στο Μαρακές ο κύριος Βέλα που είναι αυτός ο οποίος ε, υποκίνησε αυτή τη ε, διάσκεψη και το Medfish Forever και τη διακήρυξη της Σόφιας και υπενθύμησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την υλοποίηση των δράσεων για τη διαχείριση των αποθεμάτων, για τη διαχείριση του κλίματος, για την διαχείριση του περιβάλλοντος, ε, την εφαρμογή της Σύμβασης της Βαρκελόνης. Επίσης, συνολικά λοιπόν για όλα αυτά τα στοιχεία και ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι δεν βρισκόμαστε εδώ απλώς γιατί έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου, έχει ξεκινήσει ε, ένας μαραθώνιος και θα χρειαστεί χρόνος. Ε, θα πρέπει να το χτίσουμε όλο αυτό βήμα-βήμα να υπάρξει αυτή η νέα διακυβέρνηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά χάρη σε αυτή την προσέγγιση όλες οι χώρες έχουν προσχωρήσει και προοδεύουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, υπήρξε επανάσταση στη Μεσόγειο σε θέματα διαχείρισης αλίας, ε, αν ε, συζητήσει κανείς ε, τώρα με τις χώρες που βρίσκονται στο Νότο, έχουν ε, πιστεί και αυτές ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Το ίδιο γίνεται και με τον Εύξηνο Πόντο. Έχουν ξεκινήσει όλες τις προσπάθειες και οι χώρες της Μεσογείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν προσπάθειες και όταν συζητούμε με τις περιφερειακές οργανώσεις υπάρχει πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος και όταν θα συζητηθεί η νέα στρατηγική το 2020, γιατί η νέα στρατηγική θα συζητηθεί με όλες τις χώρες της Μεσογείου το 2020, θα ε, εγκριθεί από εκεί και πέρα για το διάστημα 2021-2025 και τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα εδώ θα είναι τα ουσιαστικά στοιχεία ότι πρέπει να ενισχυθούν τα επιστημονικά στοιχεία, πάντα αυτό, να υπάρχουν πολυετή σχέδια για όλα τα είδη, ε, το 100% των εμβληματικών ειδών, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα ε, δράσης για τη μικρή κλιμακασαλία, γιατί είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας στη Μεσόγειο, θα να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας, να ενισχύσουμε τις χώρες μέλη και να ασχίσουμε και τον οργανισμό για να μπορέσει να συντονίσει τα πράγματα και να υπάρχουν και κατάλληλες ικανότητες και δυνατότητες γιατί πάντα δεν έχουμε αρκετέ δυνατότητε και πρέπει να ενισχύουμε τις δυνατότητέ μας στην Αλία, να ενισχύσουμε και το περιβαλλοντικό σε θέμα. Θα επανέλθει στο θέμα αυτό η συνάδελφο, αλλά υπάρχουν κάποιες προσπάθειες οι οποίες συμφωνήθηκαν. Υπήρχε και μια επιτυχία γιατί είχαμε μια ε, περιοχή προστατευόμενη στην Αδριατική θάλασσα, στο Αδριατικό πέλαγος, και αυτό μας επιτρέπει να μπορέσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα ε, βαθύ ήβια ήδη και να μπορέσουμε να έχουμε κάποια μέτρα για τα θέματα αυτά στην Αδριατική θάλασσα και ε, έτσι ε, ξεκινούν σιγά σιγά να υλοποιούνται κάποια μέτρα στη Μεσόγειο επί τη βάση μελετών, επί τη βάση επιστημονικών αναλύσεων Αντιστοίχως ε, το πρόβλημα του κλίματος. Οι επιστήμονες ε, στο φόρουμ επεσήμαμαν ότι το 2100 αν υπήρχε αύξηση Κατά 4 βαθμούς ε, Κελσίου στη θερμοκρασία θα έχουμε 30% των ειδών που θα φύγουν από τη Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι δείκτες ε, και αυτό προσπαθούμε τώρα να καταρτήσουμε για τις συνέπειες του κλίματος ε, στα διάφορα είδη. Όσον αφορά τα χωροκατακτητικά είδη, υπάρχουν είδη τα οποία πέρασαν τη διόργα του ΣΟΕ και έφτασαν στη Μεσόγειο. Υπάρχει για παράδειγμα το λεοντόψαρα. Ε, η ε, ένα ε, ε, είδος... Cette nouvelle stratégie permettra justement ο Στράκο, ένα γαστερόπεδο το οποίο και αυτό βρέθηκε ξαφνικά στη Μεσόγειο και πρέπει κάπως να συνεχιστεί το θέμα της διακυβέρνησης. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια για το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Το 2019 θα συνεδριάσει η GFCM, θα έχουμε την ετήσια συνεδρίαση, η οποία θα ε, είναι αφιερωμένη στην έγκριση των νέων μέτρων διαχείρισης βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Προς το παρόν υπάρχουν κάποια μέτρα βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για να βοηθήσουμε την χνηλωσιμότητα, κάποια μέτρα για την Αδριατική. Πρέπει να υπάρχει ένα ε, σχέδιο με κάποια τεχνικά μέτρα και διατήρηση ε, κάποιων ε, ειδών. Θα πρέπει επίσης ε, να δούμε τι γίνεται. donc, il conviendra de mettre en place des mesures telles que la να δούμε τι γίνεται με την τσιπούρα. Επίσης υπάρχει το καλκάνι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τα τάκ και τις ποσοστώσεις, αλλά και συστήματα χνηλασιμότητας και για το καλκάνι. το μεγάλο πρόβλημα της λαθρέας και παράνομης και άναρχης αλίας ε, είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα για το καλκάνι και για το κόκκινο κοράλι που είναι ε, εμβληματικά είδη του ευξηνού πόντου και της Μεσοχείου. Υπάρχει και η Επιτροπή Εφαρμογής ε, η οποία καθόρισε ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν διαφάνεια στις συμφωνίες της Αλίας στη Μεσόγειο αλλά επίσης και κατηγοριοποίηση ε, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το γεγονός ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον κατάλογο των σκαφών ε, που είναι, ε, ασκούν παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία, ε, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση ακόμα με τα κράτη-μέλη, είναι υποσυζήτηση ακόμα και με τα αντιπροσωπευτικά όργανα, όπως για παράδειγμα το ΜΕΝΤΑΚ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ένα σύνολο προτάσεων και υπάρχει και η στρατηγική που θα εγκριθεί το 2020 και μια υπουργική διάσκεψη για τη διακήρυξη της Σόφιας για τον Εύξηνο Πόντο. Το 2021 θα έχουμε και πάλι ένα φόρουμ αλληλείας με όλους τους επιστήμονες για να αξιολογήσουμε την κατάσταση των αποθεμάτων, καθώς επίσης και όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και προβλέπεται και ένα συμπόσιο, συμπόσιο για το κόκκινο κοράλι και ε, αναθεώρηση της εφαρμογής της ε, διακήρυξης Medfish Forever. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ε, οδήγησαν σε κάποια δραστηριότητα. Ε, η μείωση των αποθεμάτων δεν είναι μοιραία, μπορούμε να την ανατρέψουμε και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσετε να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι ο στόχος ε, της ε, ε κοινή αλληλευτικής πολιτικής να έχουμε τα στόκ σε ένα διαχειρίσιμο MSY. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. thank you, Lane. that was... Ευχαριστούμε κυρία Λέιν. Ευρύτατη η παρουσίασή σας και σίγουρα μας προσφέρει κάποια ελπίδα. Δείχνει ότι η Κομισιόν προσπαθεί όντως να λύσει κάποια προβλήματα. Ε, δεν ξέρω αν θέλουν τα μέλη να θέσουν ερωτήσει. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ε, μιλήσατε, κάτι για τα επίπεδα, μιλήσατε για τα επίπεδα της βιομάζας στην προηγούμενη διαφάνεια. Είπατε ότι υπάρχει μια μικρή ε, αύξηση. Πώς υπάρχει μικρή αύξηση όταν έχουμε τόσο μεγάλη υπεραλίευση την οποία μας καταδείξατε στις προηγούμενες ε, Πώ γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Και άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχει πραγματικά σημαντική υπεραλίευση. Ε, ο... Ο γάδος ε, είναι ένα από τα ψάρια που υπεραλίευεται. Και πέραν της παρουσίασής σας, είπατε ότι πρέπει να κάνουμε ένα κβαντικό άλμα ότι είναι ζωτική σημασία. Ε, είναι μια απλή ελπίδα αυτό ή έχετε κάποια στοιχεία ρεαλιστικά. Έχετε δηλαδή, ε, έχουμε δυνατότητα να συμφωνήσουν και οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο για το βαθμό στον οποίο πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη θετική τάση, ε, συμμετείχαμε πριν από λίγο σε μια συνεδρίαση για τον εύξηνο πόντο της ε, Επιστημονικής Επιτροπής για τον εύξηνο πόντο και διαπιστώσαμε ότι ο δείκτης FMSY είναι στο 2,2%, υψηλότερος δηλαδή από το FMSY, αλλά παρατηρούμε αύξηση της βιομάζας, είναι γεγονός. Υπάρχει μια θετική τάση ανάπτυξης της βιομάζας, είναι διαπιστωμένο ε, επιστημονικά και παρατηρήσαμε την ίδια τάση και για άλλα αποθέματα. Άρα οι επιστήμονες μας δίνουν ελπίδα και δείχνουν ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον εύξηνο πόντο και σε άλλα αποθέματα έχουν ε, θετικό αντίκτυπο. Παρατηρήσαμε το, ίδιο για το Μερλούκιο, ο οποίος ε, αποτελεί αντικείμενο υπεραλίευσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια θετική τάση, αυξάνονται τα μεγέθη. Ξέρετε ότι το μέγεθος είναι μια θετική ένδειξη και στις εκφορτώσεις βλέπουμε αυξημένα μεγέθη, η βιομάζα είναι επίσης αυξημένη, άρα για μένα αυτή η αντίληψη δεν είναι 100% αισιόδοξη, αλλά δίνει θετικές ενδείξεις. Ε, αυτό συγκρατώ. Θα σας ε, σταματήσω, παρακαλώ. Για μένα και ίσως και για άλλα μέλη θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια βασικά πράγματα για την αλία. Πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Ε, Πολιτική αλίας για αρχάριους. Κάντε μια ε, μικρή παρουσίαση παρακαλώ. Για μένα και τους υπόλοιπους. <laughs> Μία απλή εξήγηση για το πώς μπορεί να αυξάνεται η βιομάζα. Ε, εδώ στο έγγραφο γίνεται αναφορά στη ποσότητα των ε, αναπαραγωγικών αποθεμάτων. Η μέση θνησιμότητα ε, και η μέση θνησιμότητα για το συγκεκριμένο απόθεμα. Τα δύο συνδέονται, αλλά ίσως κάποιες φορές ε, αυξάνεται η βιομάζα γιατί αλλιεύονται λιγότερα τα ενήλικα ψάρια. Και κάτι άλλο, ο αριθμός που έδωσε η κυρία Ελενέ είναι ένας μέσος όρος. Ε, αφορά περίπου 50 αποθέματα. Άρα τα στοιχεία που έδωσε η συνάδελφος αφορά έναν μέσο όρο για αυτά τα αποθέματα. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Και για να ε, απαντήσω στις ερωτήσεις σας, σε ό,τι αφορά την ε, υπεριαλίευση του μερλούκιου. Ε, ελήφθη η εξής απόφαση να ε, υλοποιηθεί ένα καθεστώς διαχείρισης της αλληλευτικής προσπάθειας. Πέρα από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, υπήρχε ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ο κλάδος, ρώντας την ε, ελπίδια διαχείρισης σε επίπεδα ε, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, επέλεξαν να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην, κοινωνική διάσταση και την μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε την αλία και δεδομένου του μεικτού του χαρακτήρα των αποθεμάτων. Εδώ Μερλούκιος ε, αντιπροσωπεύει ένα ε, μέρος των αποθεμάτων, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη. Όταν αλλιεύει κανείς ε, Μερλούκιο, αλλιεύει και γαρίδες, καθώς και άλλα είδη. Άρα είναι ιδιαίτερα μεικτή η αλλία σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό χρειάζεται μια τέτοια προσέγγιση, όπως σας είπα, γιατί ήταν απαραίτητη μια του κλάδου προκειμένου να εφαρμοστούν κατάλληλοι μηχανισμοί. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αντίθετα με τη Βαλτική και τον Ατλαντικό, εδώ έχουμε αλληλεία μικρής ε, κλίμακας με πάρα πολλά μικρά σκάφη. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το στόλο με κατάλληλα εργαλεία. Στη Μεσόγειο δεν χρησιμοποιούμε τις ε, ποσοστώσεις, αλλά τον αριθμό ημερών αλίας. Γι' αυτό ε, υλοποιήθηκε ένα σχέδιο με βάση τη διαχείριση της αλλιευτικής προσπάθειας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσουμε την μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα αυτά τα αποθέματα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα το φτάσουμε αυτό το επίπεδο, γιατί θα λάβουμε υπόψη όλα τα αποθέματα γιατί αυτό το σχέδιο αφορά όλα τα αλληλευτικά σκάφη, άρα είναι πολύ πιο γενική η προσέγγιση, προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της αλίας μικρής ε, κλίμακας, ε, στις μικρές ε, ποσότητες και τα είδη που αλλιεύονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτιμήσαμε αυτή την προσέγγιση, γιατί ε, ταιριάζει καλύτερα. Συζητήσαμε εκτενώς με τους επιστήμονες για το ποιο εργαλείο θα ήταν καταλληλότερο και καταλήξαμε στο σε αυτό το συμπέρασμα και καταρτήσαμε αυτό το χάρτη με που βασίζεται ε, στην διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας και στην ε, απαγόρευση της αλληλείας σε κάποιες ε, ζώνες προκειμένου να προστατευτούν οι γόνοι και τα αναπαραγωγικά αποθέματα. Για να προστατεύσουμε το μερλούκιο πρέπει να προστατεύσουμε και τους γόνους και τα αναπαραγωγικά αποθέματα. Στη Μεσόγειο λοιπόν η ε, σημαντικά εργαλεία είναι οι ε, ζώνες απαγόρευσης και η διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας. Γι' αυτό κάναμε αυτή την επιλογή και πιστεύω ότι θα φανούν σύντομα τα αποτελέσματα και θα ε, δούμε ότι μπορούν να αποκατασταθούν με κατάλληλο τρόπο τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τη Βαλερή. Ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για να γνωρίζουμε την κατάσταση της Μεσογείου και του Ευξήνου Πόντου. Στην περίπτωση του Ευξήνου Πόντου θα ήθελα να επισημάνω για να τα ακούσω και η Επιτροπή ότι ως πολιτική ομάδα η ομάδα μου αποφάσισε το επόμενο εξάμεινο να επικεντρωθεί στον εύξηνο πόντο. Θέλουμε να κάνουμε και μία ε, αποστολή, να υπάρξει και μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, για να μπορέσουμε να ε, εστιάσουμε στη συγκεκριμένη ανησυχία που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι αιτιολογημένο να κάνουμε κάποια πράγματα. Και η ομάδα μου θα ήθελε να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή ε, κάτι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του ευξήνου πόντου. Όσον αφορά την περίπτωση της Μεσογείου, ε, είναι σίγουρα ανησυχητική η κατάσταση ε, από αυτά που αντανακλώνται εδώ. Είναι λογικό ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Νομίζω ότι το σχέδιο που εγκρίναμε στο τέλος της προηγούμενης θητείας για τη Δυτική Μεσόγειο είναι στο σωστό δρόμο. Ήταν πολύ δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Ε, βασίζεται στην αλληλευτική προσπάθεια και ο στόχος είναι να έχουμε μία κατά 40% και θεωρώ ότι είναι στη σωστή άγουσα, αλλά είναι μόλις η αρχή. Υπάρχουν και άλλες περιοχές της Μεσογείου, δεν είναι μόνο η Δυτική και θα ήθελα να ρωτήσω τη Βαλερή αν και από ό,τι αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι η κατάσταση είναι προσωρινή και ότι αλλάζουμε επίτροπο και χαρτοφυλάκιο μπορεί να επηρεάσει και τα πράγματα. Θα ήθελα να ξέρω λίγο τι προγραμματισμό έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, υπόλοιπη Μεσόγειο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης, είναι ένα πρώτο βήμα και όπως είπε ο Πρόεδρος είναι και ε, δέσμευση των χωρών να ε, επιληθεί το πρόβλημα της υπεραλίευση. Και πρέπει όμως να είμαστε και Υπάρχει δέσμευση τη Ισπανίας, τη Ιταλία και τη Γαλλία για να γίνει διαχείριση. Υπάρχουν και άλλες περιοχές όμως, η Αδριατική, άλλες περιοχές της Μεσογείου και θα ήθελα να ξέρω τι προγραμματισμός υπάρχει για τις υπόλοιπε περιοχές. Και επίσης θα ήθελα, διότι δεν έχω καταλάβει ε, ακριβώς ε, τι προγραμματίζουμε ε, για το μέλλον. Η Μεσόγειος ε, όπως είπε και η Βαλερή, μπορεί να ήταν λίγο καθυστερημένη η παρέμβαση, αλλά όπως ε, είπε και η ίδια, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στη Μεσόγειο, τις οποίες γνωρίζουμε και θεωρώ ότι η αρχή έγινε με αυτό το σχέδιο διαχείρισης και είναι η πλέον κατάλληλη άγουσα για να ξεκινήσουμε. Υπάρχει επίσης μια πράξη κατεξουσιοδότηση ε, και αυτά είναι στο σωστό δρόμο. Ε, πέραν όμως το προγραμματισμό για την υπόλοιπη Μεσόγειο, θα ήθελα να ξέρω επίσης γιατί με 40 εθνικά σχέδια διαχείρισης συνεχίζουμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Ακόμα και η χώρα μου, το λέω. Όλες οι χώρες μας έκαναν εθνικά σχέδια διαχείρισης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια κάκιστη κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλύτερο να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείριση, ε, το οποίο θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικά, διότι τα εθνικά σχέδια διαχείριση ε, φαίνεται να είναι λίγο αποτελεσματικά. Τι μπορεί να μου πει η Βαλερή, γιατί αυτά τα 40 σχέδια διαχείριση δεν μας δώσαν ε, έστω ένα ελάχιστο αποτέλεσμα. Είναι πολύ ανησυχητικό γιατί υπήρξαν πάρα πολλές δράσεις και θα ήθελα να ξέρω τουλάχιστον ποια είναι η εκτίμησή τη και γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε εδώ. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι έχουμε μπει πλέον στο σωστό δρόμο και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Ε, είναι αυτό το οποίο επιτάσσει η κοινή ελευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Mr. Sullivan. Σάλιβαν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, μιλούμε για την κατάσταση στον Αξινοπόντο και στην ε, Μεσόγειο και από ό,τι ακούω από την Κομισιόν υπάρχει 87% των αποθεμάτων που υπεραλλιεύονται. Ε, είναι ιδιαίτερο υψηλό το ποσοστό αυτό. Τον, ε, Σεπτέμβριο, τον Δεκέμβριο του 2018 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ε, για το ε, πολιτές, σχέδιο για την βαθύ διαλύεια. Παρά όμως τα πολύ σημαντικά επιχειρήματα για τους ελέγχους κτλ. Το τελικό κείμενο λέει ότι την, την θα την θα την... η αλία θα τύχει διαχείριση μέσω ε, περιορισμού της προσπάθειας. Για συγκεκριμένε ε, περιοχές μάλιστα πρέπει να μειωθεί η αλληλευτική προσπάθεια κατά 10% σε σχέση με την ε, βασική γραμμή που έχουμε. Πριν από 9 μήνε το είπαμε αυτό. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή τη για την επιστοποίηση των, ισχύω των κινητήρων που είναι ένα σημαντικό για την, θέμα για, την, για το καθεστώ διαχείριση τη ε, προσπάθεια. και λέμε, μιλούμε για το 51% των πιστοποιημένων σκαφών ε, ε, η ισχύς, τους, η του κινητήρα τους ξεπερνά την, ε, ε, το δεδομένο που έπρεπε να τηρείται. Και μάλιστα το, τα, οι περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνονται στην, στην Μεσόγειο, στον κόλπο της Λιών, με τα περισσότερα, οι περισσότερες περιπτώσεις να είναι τράτες. Οι υπολογισμοί για την αλληλευτική δραστηριότητα και το σχετικό σύστημα ήταν λανθασμένο σε μεγάλο βαθμό. Οπότε το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι θα κάνετε να, για να αποτρέψετε να υπολογίζετε η ε, αληφτική προσπάθεια και η ισχύ των κινητήρων των σκαφών ε, με τον λανθασμένο τρόπο που γίνεται τώρα. Πώς μπορείτε να επιστοποιήσετε ή να αλλάξετε την κατάσταση έτσι ώστε η προσπάθεια να υπολογίζεται σωστά. Και μετά το άλλο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτείνει το υιοθετηθέν σχέδιο διαχείρισης ε, να βελτιώσει την κατάσταση για τα υπεραλλιευόμενα είδη, αν οι υπολογισμοί που γίνονται δεν αντικατοπτρίζουν το σύστημα και την προσπάθεια αλληλείας ε, που υπάρχει τώρα. Καταλαβαίνω, Πρόεδρε, ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό, αλλά ε, αν θα μπορούσε τουλάχιστον η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν και ασυνέπειες στα δεδομένα που έχουμε, καλό θα ήταν. Ευχαριστώ. Άλλος ένας ομιλητής, άλλη μία μάλλον ομιλήτρια. Χωρίς μικρόφωνο, για άλλο σημείο ήθελε η κυρία να μιλήσει. όχι απλώς... Ε, Είπα μήπω θέλατε να κάνετε κάποιο να δημιουργήσετε διπλωματικό επεισόδιο, γιατί θέλατε να μας πείτε αν ε, θα είναι 200 μίλια μακριά από το Γιβραλτάρ η, η ζώνη σας, ε, αν γίνει τελικό στο Brexit ή όχι. Λοιπόν, πάμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πολλά τα θέματα. Εγώ μίλησα για, την, ε, για το πώς θα εξοικειωθούν με το σύστημα αυτό τα κράτη-μέλη. Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η προοπτική που έχετε των 10 ετών και το σχετικό σχέδιο. Μετά, η κυρία Γκιλέρα έθιξε σε διάφορα θέματα. Άλλα διαχειριστικά πλένα, πλένα σχέδια και επίσης το θέμα της εφαρμογής. Πόσες από τις πολιτικές, ας πούμε, εφαρμόζει η Ιταλία. Πόσες μεσογειακές χώρες εφαρμόζουν την απαγόρευση και την πώληση μικρών ηχθείων Θυμά, θυμάμαι η Μαρία Δαμανάκη όταν ήταν επίτροπος έφυγε το θέμα αυτό. Ακόμα και στα δικά μας τα ψαράδικα βλέπω να πουλούνται ψάρια που δεν πρέπει να πουλούνται. Ακόμα εκεί είναι αυτά τα ψάρια. Μετά το θέμα της πιστοποίησης των κινητήρων. Και πάλι ερχόμαστε στο θέμα της ελευτικής προσπάθειας στο σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, είπαμε, το MSY μέχρι... Εντάξει, πρέπει να επιτύχουμε το MSY μέχρι το 2025 μέσω της μείωσης της ελευτικής προσπάθειας μέχρι, με μείωση 15%. Να μειώσουμε δηλαδή τα πόσα ψάρια μπορεί να πιάσει ένα σκάφος που βγαίνει να ψαρέψει. Το είχε πει και ο κύριος Βιαμών το πρωί. Οπότε μας εξηγήσατε για 40 λεπτά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το θέμα είναι τα κράτη-μέλη κάνουν το δικό τους καθήκον από τη δική τους τη μεριά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλα τα θέματα που τέθηκαν είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα συζητάμε επί μονίμου βάσεως με τις ε, χώρες της Νότιας Όχθης και άλλες χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Ε, πράγματι, στη Μεσόγειο το πρόβλημα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων. Είναι ένα από τα θέματα, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη Μεσόγειο. Ε, είναι θέμα ιστορικού χαρακτήρα. Πράγματι υπήρχε πρόβλημα εφαρμογής, αλλά όπως σας είπα δεν είναι μοιραίο. Το 2006 είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον τόνο. Η, η κατάσταση ήταν ε, καταστροφική. Υπήρχε μια ε, υπερικανότητα, υπεραλίευση σε ιστορικά επίπεδα, τεράστιες υποσότητες του, τόνου στις αγορές. Τι συνέβη. Ε, Πιστοποιήσαμε με, εξαιτίας των αντιδράσεων των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και το 2006 εφαρμόσαμε ένα σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων του τόνου με την ανάλογη προσαρμογή της αλληλευτικής προσπάθειας προβλέπονταν και κάποια μέτρα ελέγχου γιατί χωρίς έλεγχο δεν πάμε πουθενά. Και ε, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος... Ε, ε, Καθορίστηκαν ε, όρια αλευμάτων, ε, μεγέθους ε, των ψαριών, των αλευμάτων και προβλέπτηκαν διαδικασίες για τον έλεγχο όλης της διαδικασίας από την αλία μέχρι την διάθεση στην αγορά. Τι συνέβη μετά από 10 χρόνια προσπαθειών δέκα χρόνια που τέθηκε σε εφαρμογή ένας έλεγχος, αναπτύχθηκαν κατάλληλα μέτρα ελέγχου, ε, αεροπλάνα, σκάφη ελέγχου, οι πολίτες, ε, κάποιοι πολίτες αποφάσισαν να μην τρώνε τόνο. Τι συνέβη λοιπόν. Άρα ε, αυτό δείχνει ότι η περιελήψη δεν είναι κάτι μοιραίο. Αυτό που κάναμε για το τόνο μπορούμε να το κάνουμε και για το ξηφία και για άλλα Ηδη. Αυτοί οι μηχανισμοί που υλοποιούνται, ε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είναι χωρίς προηγούμενο στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μηχανισμούς ελέγχου και επιθεώρησης σε όλη τη Μεσόγειο, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα καλύπτεται όλη η Μεσογειακή λεκάνη από τα μέτρα ελέγχου και επιθεώρησης. Η υπηρεσία μας, η υπηρεσία του Βίγκου, θα συντονίζει τα μέτρα ελέγχου των κρατών μελών αλλά και των τρίτων χωρών. Αυτό είναι σημαντικό σήμερα. Ε, πείσαμε τις άλλες τρίτες χώρες να ε, εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου. Η Τινησία, για παράδειγμα, προχώρησε στην πρόσληψη 70 επιθερητών, ενώ είχαν παγώσει οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων και το δέχτηκε αυτό η ε, Τινησία ε, εξαιτίας της πίεσης που δέχτηκε από την Medfish Forever. Δύο σκάφη επιθεώρησης ε, αγοράστηκαν, ε, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί όπως είπατε υπάρχει το θέμα των ε, βαθών υδάτων στην Μεσόγειο. Η Τινησία λοιπόν είναι το τέλειο παράδειγμα που παρά τα σημερινά πολιτικά προβλήματα προσέλαβε 70 επιθεωρητές οι οποίοι συμμετείχαν σε διετή εντατική ε, κατάρτιση ε, υπό την αιγίδα της υπηρεσία μας. Ε, η Τινεσία απέκτησε συστήματα ελέγχου τύπου VMF με κάλυψη της τάξης του 80% των τινησικών σκαφών. Η Τινησία λοιπόν θα μπορεί να έχει ένα όλο που θα συμμετέχει στις προσπάθειες ελέγχου. Είπατε, υπάρχουν προβλήματα. Η Λιβύη έχει προβλήματα, αλλά ε, ε, συμμετέχουν οι, ε, οι αρχές της Λιβύης στην όλη προσπάθεια. Έρχονται επιθεωρητές από τη Λιβύη, συζητάμε μαζί τους, συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια. Οι Αιγύπτιοι επίσης έχουν δυστυχώς πρόβλημα με την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Ε, οι ε, Αιγυπτιακές αρχές ε, έχουν αρχίσει να συμμετέχουν στις προσπάθειες ελέγχου στη Μεσόγειο. Στέλνουν επιθεωρητές και συμμετέχουν στις συναντήσεις. Σήμερα καλύψαμε όλα τα ύδατα στην Αδριατική, δυτικά, ανατολικά, στον Εύξηνο Πόντο όλες οι επιθεωρήσεις με σκάφη και με ε, αεροπλάνα επιτρέπουν την, ε, τον εντοπισμό παράνομων και λαθρέων ε, δραστηριοτήτων, ε, μεταδίδονται οι σχετικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνουμε αυτές πληροφορίες, τις στέλνουμε κατευθείαν στα κράτη σημαία και ρωτάμε τι μέτρα προβλέπουν στη συνέχεια, τι διοκτικά μέτρα. Ε, αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή. Ε, αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με τη ΦΑΟ, ε, κάνουμε μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων παράνομης λαθρέας και άναρχης ε, αλίας. Οι χώρες όμως συνεργάζονται εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου των εκφορτώσεων, χρειάζεται βέβαια χρόνος, γίνονται όμως προσπάθειες οι χώρες χρειάζονται ε, ε, βοήθεια, υποστήριξη για την απόκτηση σκαφών, την ευαισθητοποίηση των αλλιέων, στην νοτροπία ε, συμμόρφωσης, προκειμένου και οι ίδιοι οι αλλοίς καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τα μέτρα διατήρησης. Φέτος διαπιστώσαμε, ανακαλύψαμε ότι στο κανάλι της Σικελίας οι αλλοίς δέχονται την παρουσία επιθερό τόνο στα σκάφη τους. Ε, τα ανοίγματα των δικτυών έχουν, ε, είναι πιο μεγάλα τώρα και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων των μέτρων που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα. Μας βοηθάει και η Frontex, ε, μας βοηθάνε και άλλες ε, υπηρεσίες και όλα αυτά ε, δείχνουν ότι η πολιτική ελέγχου, η νοτροπία ελέγχου στην ε, Μεσόγειο αλλάζει, εξελίσσεται. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες, στοιχεία, Έχουμε ε, ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν προκειμένου οι χώρες του έξινου Πόντου και της Νότιας Όχθης Μεσογείου να ε, καταβάλουν προσπάθειες. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας ε, Αγγιλέρα, πρέπει πράγματι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να εφαρμοστούν σχέδια διαχείρισης σε όλη τη Μεσόγειο. Υπάρχει μια επίσημη δέσμευση στα πλαίσια της Medfish Forever για την κάλυψη συγκεκριμένου του, των αποθεμάτων. Σε κάθε συνάντηση ε, εφαρμόζουμε σχέδια σε ό,τι αφορά την Αδριατική. Έχουμε υλοποιήσει ένα σύστημα συλλογής δεδομένων και ε, βάσιμων επιστημονικών ε, γνωμών. Μόλις έχουμε λάβει έτοιμα ε, από την Επιστημονική Επιτροπή της Αδριατικής που να λάβουμε μέτρα προκειμένου να να υπάρξει μια διαχείριση της ε, αλληλευτικής ε, προσπάθειας, ε, να ληφθούν μέτρα ελεγκτικά και πρέπει να δούμε σε, τι, σε ποιο επίπεδο πρέπει να γίνει η διαχείριση των αποθεμάτων στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο του GFCM. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό ακόμα. Θα ληφθεί μια απόφαση στο μέλλον. Προς το παρόν επήγει να υλοποιηθεί ένας ε, χάρτης για τη διαχείριση των ε, βενθοπαλλαγικών ε, αποθεμάτων στην Αδριατική. Στους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια θα καταρτιστούν χάρτες για όλα τα αποθέματα που είναι, αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης και έχουν κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την υπεραλίευση. Ε, στη ε, δυτικά πράγματι ε, όπως είπε η συνάδελφος, έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα ελέγχου της αλλιευτικής προσπάθειας. Αυτό το σύστημα υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετήθηκε τον ε, περασμένο Αύγουστο. Προβλέπονται συγκεκριμένες ε, ποσοστώσεις, οι οποίες θα ε, συζητηθούν το Δεκέμβριο όταν καθοριστούν οι αλληλευτικές δυνατότητες. Οι ποσοστώσεις αυτές θα εκφράζονται υπό τη μορφή ημερών αλίας, ε, και με βάση τους υπολογισμούς των κρατών ε, μελών για την αλληλευτική προσπάθεια για την περίοδο 2015-2017 και προβλέπεται μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας της τάξης του 10%. Ε, συνολική προσπάθεια μείωση προβλέπεται στα 40% τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Υλοποίησαμε λοιπόν ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάθε αλλιέας θα πρέπει να ε, καταγράφει τον αριθμό ημερών αλλιείας, τις αλλιευτικές ζώνες, ε, αυτές οι ε, πληροφορίες θα μεταφέρονται ή ε, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο στο κράτος σημαία. Σε μηνιαία βάση το κράτος σημαία θα πρέπει να μεταδίδει αυτά τα στοιχεία στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να ενημερώνει επίσης αν έχουν επιτευχθεί ή ε, ποσοστώσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν θα υπάρχει ένα καθεστώς ελεγχόμενης αλληλευτικής προσπάθειας και αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή της αλληλευτικής προσπάθειας και το περιορισμό της υπεραλίευσης στην περιοχή. Και κάτι πολύ σημαντικό θα περιορίσουμε τον αριθμό ωρών για κάθε ημέρα αλίας, 15 ώρες αλίας κάθε μέρα και 5 μέρες αλίας ανά εβδομάδα. Άρα με μαθηματικό τρόπο θα μειωθεί η αλλιευτική προσπάθεια και κάτι άλλο πολύ σημαντικό θα επεκτείνουμε τον έλεγχο και σε αυτή την ε, περιοχή. Η υπηρεσία μας λοιπόν θα μπορεί να ε, προβαίνει στους ελέγχους και να τους ε, συντονίζει. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα έχει καθοριστεί ανάλογα με τα αποθέματα Πράγματι όμως η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγξει το σύνολο των μηχανισμών που προβλέπονται ε, από τον ε, ε, κανονισμό. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μπορεί μαζί με τα κράτη-μέλη να ε, γνωρίζει την πραγματική κατάσταση των ε, στόλων και να προβαίνει στις κατάλληλες προσαρμογές. Εγώ ε, δεν είμαι ίδια στην Επιτροπή, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα αν τυχόν συγκεκριμένη παρατηρηθεί η υπέρβαση της συγκεκριμένης ισχύω των στόλων. Ε, εδώ και κάποιο καιρό ε, αξιολογούμε αυτά τα ανώτατα όρια και τον έλεγχό τους είναι δύσκολο να ελεγχθεί η κινητική ισχύ των ε, στόλων. Είναι δαπανηρό, αλλά είμαι σίγου... χαίρομαι πολύ που η Επιτροπή έχει λάβει αυτά τα μέτρα. Συμφωνούμε μαζί σας, κυρία Λέν. Αλλά αυτό που είπε η συνάδελφος είναι ότι συχνά ε, αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονται και συνεχίζονται κάποιες ε, παράνομες ε, δραστηριότητες. Όπως σας έλεγα, η Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της και ε, με βάση τις αδυναμίες που θα διαπιστωθούν θα ε, αναλάβει και την απαραίτητη δράση. Θα επικοινωνήσει με τα κράτη-μέλη προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα ε, μέτρα για την τήρηση των ορίων της ισχύω των στόλων. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ ε, τολμηρό. Οι, τα κράτη-μέλη έχουν ε, υποχρέωση να πιστοποιούν την ισχύ των ε, σκαφών. τώρα η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη, όπως και για όλα τα μέτρα που δεν εφαρμόζονται, θα τα καλέσει λοιπόν να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα διαφορετικά. Θα θα αντιμετωπίσουν ε, ε, κυρώσεις, τις κυρώσεις που προβλέπονται. Η κυρία Αγγιλέρα ρώτησε για το τι προβλέπετε για την υπόλοιπη ε, Μεσόγειο, τις ε, υπόλοιπες περιοχές, έτσι δεν είπατε κυρία Αγγιλέρα. Ρωτήσατε στην Κομισιόν τι θα γίνει στη συνέχεια. Ναι, αλλά απάντησε η κυρία της Επιτροπές. Αναφέρθηκε στο προγραμματισμό της Αδυρατικής και όλο τον προγραμματισμό που προβλέπεται στις υπόλοιπες περιοχές. Ναι, ναι, τα ανέφερα. Αυτό που ρώτησα επίσης είναι τι έγινε, διότι με τόσα εθνικά σχέδια ε, δεν είχαμε σχεδόν καθόλου επιτυχία. Προφανώς ε, με αυτό που είπε η Βαλερή είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν παρκώς τα μέτρα. Είναι σαφές νομίζω με αυτά που είπε η Βαλερή. Ναι, αλλά θέλω να κλείσω τον κατάλογο των ε, αγορητών. Μία σύντομη ερώτηση πριν ε, κλείσω τον κατάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου για τη θάλασσα και τις ακτές, ε, του Υπουργείου που ήταν αρμόδιο για τις θάλασσες, ε, για ένα χρόνο ε, εργάστηκα σε ένα πρόγραμμα διάσωσης της Μεσογείου. Συγγνώμη, ήρθα όταν είχε ήδη προχωρήσει η συζήτηση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, διότι μας ενδιαφέρει με ποιες συνθήκες ε, θα προφυλάξουμε τη Μεσόγειο, γιατί ε, υπάρχει πίεση προς τους ε, αλείς, αλλά υπάρχει και πίεση λόγω της ρήπανσης της Μεσογείου και αυτή είναι και μία από τις ερωτήσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για τις πετρελοκυλήρες και την ε, μείωση της ε, ε, διάχυτης ρήπανσης και της μείωσης της ρήπανσης από τα πλαστικά. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον καλύπτει τις εργασίες στην Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για τα θέματα αυτά και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε η Μεσόγειος να μην είναι τόσο γεμάτη ρήπανση. Εγώ συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα με πολλούς ε, παράγοντες ε, για την ε, Μεσόγειο και η μείωση των σημείων που έχουν πληγεί από πετρελοκυλίδες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, ως Ευρωβουλευτή, την προηγούμενη εβδομάδα πήγα στην Τινησία, Ισία, ε, στο Φόρουμ της Θάλασσας και η Ισία δραστηριοποιείται πάρα πολύ για την ε, γαλάζια οικονομία και την διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτων οικοσύστηματων. Πρόκειται για μια χώρα η οποία ε, πραγματικά δεσμεύτηκε από αυτού και ζητούν απλώ συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και η ερώτησή μου αφορά τη μείωση της ρήπανσης λοιπόν και πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το θέμα αυτό ε, και τι συνεργασία υπάρχει μεταξύ των διαφορών γενικών διευθύνσεων. Ευχαριστώ. Ρήπανση και εθνικά σχέδια διαχείρισης, εφαρμογή κλπ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια, συγγνώμη δεν απάντησα. Υπάρχουν 40 εθνικά σχέδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να φροντίσει αυτά τα εθνικά σχέδια να αναπροσαρμοστούν βάσει των στόχων της κοινή ελευθερική πολιτικής, δηλαδή του MSY. Στείλαμε τα, τα προγράμματα. Αν θέλετε, τα περάσαμε από ένα πλυντήριο, τα στείλαμε και στον αρμόδιο οργανισμό του ΣΤΕΚΦ ε, για να μας ε, δώσει μια γνωμοδότηση και περιμένουμε τη γνωμοδότηση για το σύνολο των σχεδίων αυτών και βάσει αυτών θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν και να διορθώσουν το ε, πρόγραμμά του. Κάποιες χώρε έκαναν ήδη πράγματα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά από τη γνωμοδότηση για το εθνικό σχέδιο τη Ιταλία μείωσε και άλλαξε το εθνικό της σχέδιο και μείωσε την αλληλευτική προσπάθεια κατά 8% ετησίω για να προσαρμόσει το εθνικό σχέδιο στις συστάσεις του οργανισμού. Αυτό το κάνουμε για όλες τις χώρες τώρα. Όλες οι χώρες λοιπόν επανεξετάζουν το σχέδιό τους και ελπίζουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα μπορέσουν να ε, επανεξετάσουν τα σχέδια και να τα διορθώσουν, αλλά Σα λέω και το καθησυχαστικό ότι οι συνάδελφοι από την Ιταλία ήδη το έκαναν και χαιρόμαστε που η Ιταλία μείωσε την αλληλευτική προσπάθεια και τα προσαρμόζουν στου στόχου τη κοινή αλληλευτικής πολιτική και του MSY. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η προσαρμογή, να δέχονται μείωση κατά 8% τη αλληλευτικής προσπάθεια στο παρόν πλαίσιο και θέλουμε να το επισημάνουμε γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όπου η Ελλάδα ε, προσάρμοσε το στόλο της. Υπήρχε ένα ε, πρόγραμμα ε, απόσυρση 700 σκαφών, δηλαδή θα διαθέτει 700 λιγότερα σκάφη για να προσαρμόσει το στόλο της. Στην Ισπανία η Ισπανική κυβέρνηση προσαρμόζει τώρα το σχέδιο αλίας για να λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις του ΣΤΕΚ Βλέπετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι τα κράτη μήλη κάνουν και αυτές προσπάθειες ε, για να επιτύχουν τους στόχους MSY. Ε, μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από τον Ατλαντικό γιατί ξεκινήσαμε αργότερα, αλλά υπάρχουν προσπάθειες και συνεχίζουν να προσπαθούν. Όσον αφορά τη δική σας την ερώτηση κυρία Σαμπό, ε, πράγματι Είμαστε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα, γιατί η Γενική Διεύθυνση Έρευνα ξεκίνησε δύο μεγάλα προγράμματα για τον αντίκτυπο τη ρήπανση ε, στα θαλάσσια είδη και τα αποθέματα τη Μεσογείου. Για κάποιε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσει ζητήσαμε συγκεκριμένε νομοδοτήσει, τι οποίε ε, ε, χρηματοδοτούμε για τον αντίκτυπο του πλαστικού για τα πελαγικά είδη και επαληθεύθηκε όντω ότι υπάρχει αντίκτυπος της ρήπανση από τα πλαστικά στην ανάπτυξη της αρδέλας. Θα είναι, είναι αρνητικός βεβαίως ο αντίκτυπος και υπάρχουν και κάποιες μελέτες εξέλιξη και για άλλα είδη πλαστικών και προχωράμε και μία μελέτη για την ηχορύπανση Ξέρω ότι είναι καινούριο, αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο έχει πραγματικές συνέπειες. Έγιναν κάποιες ε, ε, μελέτες και θα γίνουν και κάποιες μελέτες στους επόμενους μήνες για την ηχορύπανση και πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη των ε, αποθεμάτων. Έγιναν κάποιες μελέτες στην Ορβηγία οι οποίες έχουν αποδείξει ότι η χορύπανση, είτε λόγω της κίνησης στη θάλασσα, είτε λόγω της, των εξορίξεων για φυσικό αέριο, υπάρχει αντίκτυπες για τα, ε, την ανάπτυξη των ειδών. Ε, στην Ανδριατική επίσης υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες μελέτες και στον Πόντο. Επομένως ε, ζητήσαμε από την Επιστημονική Επιτροπή να λάβει υπόψη τα θέματα αυτά και να υπάρξουν κάποιοι δείκτες για την αξιολόγηση των αποθεμάτων για να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία από ό,τι φαίνεται ε, έχουν συνέπειες για τα αποθέματα. Θεωρώ ότι η ολιστική προσέγγιση, η προσέγγιση ως προς το οικοσύστημα οδεύει προς την κατεύθυνση που αναζητούμε και ελπίζω και το φόρουμ και ελπίζω να μπορέσετε να συμμετάσχετε και στο επόμενο επιστημονικό φόρουμ που θα χρηματοδοτήσουμε και θα υλοποιήσουμε με την ε, ε, GFCM ε, διότι θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρες για να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα αποθέματα. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Well, thank you very Ευχαριστούμε. Ε, πείσατε πολλούς από εμά που ότι δεν είναι νοθροί η Κομισιόν ε, για τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακούσει στο, ότι στο Βόρειο Ατλαντικό υπάρχουν 81 ε, αποθέματα και μόλις ε, ε, ελάχιστα από αυτά, 59 ε, έχουν φτάσει το επίπεδο FMSY στην Μεσόγειο τι γίνεται, θα έρχεστε κάθε χρόνο και θα μας λέτε ότι τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται σε σχέση με έναν μετρήσιμο στόχο. how are we going to be able to assess... Πώς θα την ε, μετρήσουμε αυτή την πρόοδο, πώς την αξιολογούμε την πρόοδο. I have a dream θα έλεγα. Θα ήθελα να έχω αυτό το όνειρο, να μπορέσω να σας πω ότι ε, συγκεκριμένος αριθμός αποθεμάτων θα βρίσκεται στα επίπεδα της μέγισης βιώσιμης απόδοσης. Ε, ξέρετε ότι στη Μεσόγειο έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες ε, διαχείρισης. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να μπορούμε να, να υπολογίσουμε το MSY. Κάποιες χώρες δεν το έχουν κάνει αυτό. Για να είναι μετρήσιμη η φιλοδοξία μας, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη γνώση των αποθεμάτων, να έχουμε περισσότερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Πιστεύω πάντως ότι όλες αυτές οι θετικές ενδείξεις που συλλέγουμε ε, δεν λένε μόνο οι επιστήμονες ότι, υπάρχουν, ότι διαπιστώνουν βελτιώσεις. Ε, είναι κάτι που θα μπορούμε να διαπιστώσουμε κάθε χρόνο. Αυτό επιθυμεί η Κομισιόν. Σας δώσω και ένα παράδειγμα. Ε, στην Αδριατική εκεί ε, αυξήθηκε η βιομάζα, αυξήθηκε το μέγεθος των ε, ψαριών, κάτι είναι πολύ ε, θετικό, πολύ θετική ένδειξη για την απαραγωγή των αποθεμάτων. Οι επιστήμονες εργάζονται πάνω σε αριθμητικά στοιχεία και τόσο για το χάρτη που υιοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, όσο και για τους υπόλοιπου ε, χάρτες, πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα έχουμε θετικές ενδείξεις. Εδώ και τρία χρόνια ε, εφαρμόζουμε αυτή τη πολιτική και μπορώ να σας πω ότι ε, υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Του χρόνου ελπίζω πως η Κομισιόν θα, μπορεί, θα μπορέσει να έρθει και να σας δώσει περισσότερα αριθμητικά στοιχεία ε, βασισμένα σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα έχουμε την ίδια αξιολόγηση που έχουμε και στην Ατλαντικό. Στον Ατλαντικό αυτά τα σχέδια άρχισαν να εφαρμόζονται ε, εδώ και ε, πριν από 10 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Και στη Μεσόγειο λοιπόν χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να φτάσουμε τα, τη μέγιστη βιώσιμη την μέγιστη βιώσιμη απόδοση που έχει οριστεί. Το 2020 προβλέπεται η υιοθέτηση σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν να υλοποιηθούν και άλλα μέσα. Ε, πάντως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ε, οι φορείς, οι αλληλείς, τα κράτη-μέλη, τα άλλα κράτη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες, όπως το διαπιστώσαμε και στο Μαρακές. Ελπίζω λοιπόν ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων και τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε με αγωνία του χρόνου. Και ευχαριστούμε βεβαίως για την παρουσίασή σας. Πολύ, περιμέ... Πολύ την θεωρήσαμε αρκετά πιο θετική από ό,τι περιμέναμε. Πάμε λοιπόν στο σημείο 10. Ε, διακυβέρνηση των ε, ε χωρών ανάκτηση των ηχθειοποθεμάτων και προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχέ. Το άρθρο 8 τη κοινή αλληλευτική πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα καταγράψουν όπου είναι δυνατόν Ποιε είναι οι περιοχές ανάκτησης ήχθη αποθεμάτων. Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτή η περιοχή ανάκτησης, αλλά ε, ήρθα σε επαφή με τον καθηγητή Κάλαν Ρόμπερτς, που είναι βιολόγο. και ρώτησα ποια είναι τα καλά παραδείγματα τέτοιων περιοχών. Η Ισπανία μου είπε καλύτερα, τις καλύτερες περιοχές έχετε μια περιοχή την, ε, η οποία έχει πολύ, μικρής, ε, πολύ μικρό δικτύπου α, α, ε, μικρής κλίμακας αλληλεία γύρω της και, και έξω από αυτή μια περιοχή βιομηχανοποιημένης αλλιεύσης. Υπάρχουν περιοχές οτοκίας εντός της, του χώρου ανάπτυ, ανάκτησης, οπότε πραγματικά κερδίζουν όλοι. Τι γίνεται λοιπόν σε σχέση με το άρθρο 8 της κοινή αλλιευτικής πολιτικής πρέπει να δούμε και μετά υπάρχει και το θέμα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που προκύπτουν ε, λόγω αρκετά σημαντικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 12% νομίζω είναι των παρακτήων περιοχών είναι προστατευόμενες ε, περιοχές, καλύπτονται δηλαδή, αλλά μόλις το 2% έχει σχέδια διαχείρισης. Οπότε το ερώτημα είναι Κάνουν τα κρατημέλη αυτό που πρέπει. Λοιπόν, ε, σίγουρα θα το σκοτώσω το όνομά σας. Η κυρία Βεγκασκέτ, ε, συγγνώμη, από την Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει, εκπρόσωπος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε φορά, η κάθε παρουσίαση που κάνω, ε, πάντα σε κάθε παρουσίαση που κάνω πάντα πρέπει να ε, προφέρω το όνομά μου. Ελπίζω σύντομα να έχουμε και το νέο Λιθουανό Επίτροπο. Σίγουρα με το αγγλικό του όνομα θα τον φωνάζουμε παρόλα αυτά. Ποιο είναι το αγγλικό του όνομα, βάση περιπτώσει. Ε, ξέρω ότι έχουμε λίγο καθυστερήσει, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπατε να κάνω εγώ τώρα μια παρουσίαση για την αλληλεία για αρχάριους, έτσι ώστε να επαναλάβουμε λίγο ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε μέσω της ε, κοινή ελευτική πολιτική και ποιε είναι οι διαδικασίε. γιατί καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα και πάντα καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε. Αν είναι πολύ εκπαιδευτική η προσέγγιση μου, δεν προσπαθώ να σας, ε, υποβι... σας υποβιβα... υποτιμήσω ότι δεν ξέρετε, απλώς προσπαθώ να τα πω λίγο απλά. Πρόεδρε, καταρχάς σας ευχαριστώ που μας, ε, μας καλέσετε να παρουσιάσουμε το σημείο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στο άρθρο 8 και στο άρθρο 11, όπως είπατε στην αρχή, καλό είναι να σημειώσουμε ότι όταν μιλούμε για αυτά τα δύο άρθρα και αυτές τις περιοχές ε, του χώρου χώρους ανάκτησης δηλαδή και τι προστατευόμενε περιοχές. Έχουμε δύο πολιτικές εδώ σχετικά. Περιβαλλοντική πολιτική και αλληλευτική πολιτική που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε ότι έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες που παρεμβαίνουν. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές είναι μεικτές, μεικτή αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη. Η αλληλευτική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ε, όπου μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει μέτρο. Οπότε είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και αυτό όταν μιλούμε για αυτές τις περιοχές, γιατί όταν κάνατε την εισαγωγή για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, είναι σημαντικό να θυμίσω ότι αυτό είναι ευθύνη κράτους μέλους και είναι βεβαίως προνόμιο των κρατών μελών να καθορίσει ποιες είναι αυτές οι περιοχές και να λάβει και τα μέτρα ε, διατήρησης των αποθεμάτων σε αυτές τις περιοχές. Στα πλαίσια τώρα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν αυτές τις ε, χώρες είτε ε, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα οικοσυστήματα ή σύμφωνα με το πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Όλα αυτά τα πλαίσια Ξέρετε ότι τα διαχειρίζονται οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Αν θέλετε τώρα να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτέ τι νομοθετικέ πράξει, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο είναι αυτή που θα σα διαφωτίσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνει η κοινή ελευτική πολιτική για να συμβάλλει σε, αυτή την, ε, σε αυτέ τι νομοθετικέ πράξει τι περιβαλλοντικέ. Εδώ είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η νέα κοινή ελευτική πολιτική, όταν άρχισε να ισχύει το 2014, συμβάλλει πολύ πιο σημαντικά στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Και κυρίως πέραν δηλαδή των βασικών αρχών του τρέχοντος, της τρέχουσας κίνησης ελευθερικής πολιτικής για την αρχή της προστασίας, τον ορίζοντα για το 2020, όλα αυτά ήδη συμβάλλουν ούτως ή άλλως στην περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά έχουμε και δύο νέα εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να επιτύχουν ε, τους στόχους αυτής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όπως είπατε και εσείς, είναι το άρθρο 8 που έχει να κάνει με, τον καθορισμό των ε, χώρων για την ανάκτηση των ε, χθιαποθεμάτων και το άρθρο 11 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα ε, συντήρησης που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να επιτυχούν τις απαιτήσει της περιβαλλοντική νομοθεσίας. Λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο, άρθρο 8. Οι περιοχέ ανάκτηση των ηχθειοποθεμάτων. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο του κυρίου Κάλλον που αναφέρατε, είναι εξαιρετικό. Άρθρο 8 λοιπόν, προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να καθορίσουν ε, τέτοιες περιοχές ανάκτησης ε, ηχθιαποθεμάτων που είναι βιολογικώς ευαίσθητες. Αυτές οι περιοχές συνήθως, μάλλον θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ε, αποδείξεις ότι έχουν συγκέντρωση ηχθείων κάτω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος και ότι είναι και χώριο τοκίας. Στις περιοχές αυτές τα κρατημέλη μπορούν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν αληφτικές δραστηριότητε. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν ποιε είναι αυτές οι περιοχές που είναι κατάλληλε. και τα μέτρα που θα προτείνουν θα πρέπει να περάσουν μέσω τη ε, διαδικασία περιφερειοποίησης. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, η πρόοδο ποια είναι τώρα μέχρι στιγμή. Δυστυχώς μικρή είναι η πρόοδος για το άρθρο 8, το ξέρετε πιστεύω. Από το 2013 δεν έχουμε καταφέρει να λάβουμε ε, μια κοινή σύσταση στα πλαίσια του άρθρου 8. Η έλλειψη προόδου μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη γνώση ό,τι αφορά την, ε, παρουσίαση ή τον έλεγχο των απειλών για τον καθορισμό αυτών των ε, βιολογικώ ευαίσθητων περιοχών. Βεβαίω συμφωνούμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα εργαλείο που μα δίνει η, ε, η νομοθεσία. Και τα κρατη είναι αυτά που πρέπει να αναλάβουν τέτοιου είδου μέτρα για να, και να κάνουν συστάσει. Αλλά το άρθρο 8 δεν είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στα πλαίσια τη εργαλειοθήκη τη ΚΑΠ για να επιτύχουμε του στόχου. Και θα ήθελα εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, τεχνικών μέτρων και του σχετικού κανονισμού που υιοθετήθηκε πρόσφατα. Πρώτη φορά υπάρχει το εργαλείο περιφερειοποίηση για τα κρατη για να υιοθετήσουν περιφερειακά μέτρα τα κρατη για να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα ή να προστατεύσουν τι ευαίσθητε περιοχέ. Οπότε βασιζόμαστε στα κρατη και πρέπει αυτά να ενισχύσουν τι προσπαθίε του και σύντομα να υποβάλουν κοινέ προτάσει για, να βελτι... για να προστατεύσουμε αυτέ τι περιοχέ. Άλλο ένα καλό παράδειγμα, όπω είπε και η Βαλερία στη δική τη παρέμβαση, είναι το πολιετές σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα προστασίας για τα χθιαποθέματα, όπου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ε, τράτα σε, πάνω από έξι ε, ναυτικά μίλια οι χώρες της ε, Μεσογείου δουλεύουν πάνω στο να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικέ επιλογές που δίνει ο χάρτης για να μπορέσουν να, προτείνουν επιπλέον δυνατότητες ε, κλεισίματος και να προστατεύσουν τα ενδιατήματα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι έτσι θα υπάρξει μείωση κατά τουλάχιστον 20% της αλίευσης των αγώνων και αυτή η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο εργαλείο που έχει η εργαλειοθήκη της ΚΑΠ, είναι το άρθρο 11, όπου έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο να παρατηρήσουμε. Να εξηγήσω λίγο γρήγορα τι είναι. Το άρθρο 11 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη, πάλι μέσω της περιφερειοποίησης, να ε, από κοινού να ε, προτείνουν μέτρα συντήρηση σε σχέση με την αλίευση ε, σε μια συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή, η οποία, όπως είπα, μπορεί να καθοριστεί δυνάμει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όπως είπα, είναι ίδια η διαδικασία, όπως με το άρθρο 8, τα κρατημέλη δηλαδή πρέπει να προτείνουν κοινέ συστάσεις και... Μετά πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα συμβουλευτικά όργανα και ύστερα υποβάλλουν την πρόταση στην Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει τρει μήνες για να υιοθετήσει ή να απορρίψει τις κοινέ αυτές τις στάσεις. Εάν η STCF μας πει ότι αυτή η συμβολή μπορεί να επιτύχει τους στόχους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τότε αυτές οι κοινέ συστάσεις μπορούν να μεταφραστούν σε κατεξουδότηση πράξη, η οποία μπορεί να υιοθετηθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων και εδώ παρεμβαίνει το Κοινοβούλιο, γιατί σε αυτές τι κατεξοδότηση πράξεις ε, θα τις μελετήσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βεβαίως και το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο έχουν δύο μήνες ή τέσσερις στη διάθεσή του για να μελετήσουν αυτέ τι καθεξοδότητε πράξει και να πούν αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Οπότε το Κοινοβούλιο, από κοινού με το Συμβούλιο, παίζει ένα σημαντικό ρόλο εδώ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι σύμφωνα με την τελευταία ε, υπόθεση στο δικαστήριο, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι τα μέτρα συντήρηση που προτείνονται σε αυτές τις κοινέ συστάσει στα πλαίσια του άρθρου 11 δεν απαιτείται από μόνες τους να επιτύχουν τους στόχους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξή του. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το σημείο και πρέπει να το θυμόμαστε. Η CFP δεν μπορεί να ε, επιτύχει μόνη τη την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία και τι απαιτήσει τη. Πρέπει να συμβάλλει ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Μετά, τι γίνεται τώρα με το που βρισκόμαστε και την πρόοδο. Όπως είπα, το άρθρο 11 έχει προχωρήσει καλύτερα από το 8. Μέχρι τώρα έχουμε λάβει 8 κοινέ συστάσεις από τα κράτη-μέλη που μεταφράστηκαν σε έξι κατεξουδότηση κανονισμού τέσσερι εκ, οποίων, εκ τώρα είναι σε ισχύ. Ένας από αυτούς ανακλήθηκε το 2015, ήταν ο, καθ, ο, του 2015 και ένας δεν πέρασε από την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οι συστάσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, κυρίως για την Βαλτική και για τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχουν ε, κοινέ συστάσεις για τη Μεσόγειο, αλλά παρόλα αυτά έχουμε άλλα εργαλεία για τη Μεσόγειο, ούτω ή άλλω, που έχουν στόχο να επιτύχουν του ίδιου στόχου. Και εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή GFCM έχει, έχει υιοθετήσει εννέα συστάσεις για να δημιουργηθούν ε, περιοχές περιορισμένης αλίας και άλλη μια επιτυχημένη ιστορία εδώ πρέπει να αναφερθεί είναι η ε, περιοχή περιορισμένης αλληλείας στην Αδριατική που ήδη έχει επιστημονικός ωφέλη για τον ε, Μερλούκιο και για τον Αστακό. Ε, είναι λοιπόν αργή η πρόοδος για το άρθρο 11, παρόλα αυτά έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία προχωρούν, είναι στην φάση της ολοκλήρωσης, αλλά παρόλα αυτά προχωρούμε αργά και περιμένουμε ότι τα πράγματα θα πάνε και λίγο πιο γρήγορα. Ε, θεωρούμε ότι η αργή αυτή πρόοδος εξηγείται και από τη δυσκολία να βρεθεί συνένεση μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων. Οπότε στη διαδικασία έχουμε βεβαίως και τη συμμετοχή των Υπουργείων Αλίας, Περιβάλλοντος, έχουμε τους Αλίες, έχουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οπότε η αργή πρόοδος δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ισόρροπη λύση που να μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλους. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Η περιφερειοποίηση επίση ε, ε, ε, ζητά πολύ μεγάλε προσπάθειες από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και καμιά φορά είναι και θέμα δυνατοτήτων των κρατών μελών. Οπότε η περιφερειοποίηση νομίζω είναι μια διαδικασία που ακόμα δημιουργείται ουσιαστικά και ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που είναι δύσκολο για τις περιφερειακές ομάδες να διαχειριστούν όσα πρέπει να διαχειριστούν. Από τη δική μας την πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενά εμπλέκεται και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όταν λέει, η όταν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Μάρε και Περιβάλλοντος επίσης. Και ενεργώς λοιπόν ε, συμμετέχουμε ώστε να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία. Συμμετέχουμε τακτικά στις διάφορες συναντήσεις που γίνονται, όπου συζητώνται οι διάφορες, τα διάφορα σχέδια κοινών συστάσεων, δίνουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να τις βελτιώσουν πριν τις ολοκληρώσουν. Πέρσι δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο καθοδήγησης ε, που έδινε στα κράτη-μέλη περισσότερες λεπτομέρειες ε, για το ποια είναι τα μέτρα συντήρησης τα οποία προβλέπονται ή πώς θα πρέπει να τα εκπονήσουν στα πλαίσια του άρθρου 11. Και επίσης έχουμε θίξει και τις ανησυχίες μας για την αργή ε, βάση που το βάλαμε στα διάφορα του ε, Συμβουλίου του Ιουνίου. Ε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερα κονδύλια, γιατί το, ΕΦΤΑ έχει, το ΕΤ θα έχει ε, κονδύλια που είναι αφοσιωμένα στην διαχείριση της βιώσιμης αλληλείας για τη βελτίωση συλλογή δεδομένων, οπότε υπάρχουν στα χέρια μας εργαλεία. Και κλείνοντα να πω ότι έχουμε τα εργαλεία και στην κοινή πολιτική. Ναι, η πρόοδος είναι αργή, από θα θέλ, πιο αργή από θα θέλαμε, αλλά από τη δική μας την πλευρά ή από την πλευρά της Κομισιόν ενεργά συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και με τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε πώς μπορούμε να τη διευκολύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί λίγο η ταχύτητα με τον καιρό και βεβαίως ευχαρίστως να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, can you uh, indicate... Εγώ ευχαριστώ. Μπορείτε να μας πείτε το feedback που έχετε από τις συναντήσεις με τα κράτη-μέλη. Είπατε ότι κάνετε συζητήσεις. Τα κράτη-μέλη τι σας λένε. Γιατί δεν ε, χρησιμοποιούν καλύτερα την ε, νομοθεσία. Γιατί είναι τόσο αργή η πρόοδος. Και επίσης, υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των ε, περιοχών, ας πούμε, ανάκτησης αποθεμάτων και των προστατευόμενων περιοχών οι νομικές βάσεις τους είναι διαφορετικές. Αλλά όπως είπα, όπου υπήρξαν τέτοιου είδους ε, περιοχές έχουν ε, δείξει ωφέλη για την αλληλεία. Αλλά παρόλα αυτά μου λένε ότι έχουμε πάνω από 3.000 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Αυτές οι περιοχές μπορούν να δηλωθούν ως τέτοιες για να προστατευτεί το οικοσύστημα και όχι τα ψάρια. Άρα είναι δυνατόν να θεωρηθούν σε πολλές περιπτώσεις ως ε, περιοχή ανάκτησης ουσιαστικά των ε, αχθιαποθεμάτων. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να δώσουμε διαφορετική κατεύθυνση στις προσπάθειές μας ώστε οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές να τύχουν καλύτερης διαχείρισης αντί να ανησυχούμε για τις περιοχές ανάκτησης των αποθεμάτων. Αν θέλετε να απαντήσετε τώρα, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ωραία, μου απαντάτε και μετά δίνουμε το λόγο στους ομιλητές. Ευχαριστώ. Για την αργή πρόοδο, τα κράτη-μέλη πάντα μας λένε το ίδιο. Ότι είναι δύσκολο να βρουν συνένεση, αν υπάρχουν διάφορα κρατημέλη γύρω από ένα τραπέζι έχουν διαφορετικά συμφέροντα, πρέπει να δουν και τη δική τους, το δικό τους κλάδο αλίας ο καθένας, τα διάφορα υπουργεία αλίας πρέπει να συμφωνήσουν. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρεθεί μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση για όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή, νομίζω, του, του κόσμου τη Ελία. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλε τι πλευρέ και αυτό είναι ο βασικό λόγο. Για το ερώτημά σα τώρα για την επικάλυψη μεταξύ των χώρων ανάκτηση και των προστατευόμενων περιοχών, Όντω, οι περιοχέ οι περιοχές προστατευόμενε μπορεί να θεωρηθούν χώροι ανάκτηση. Θα μπορούσαν φυσικά να βελτιωθούν ε, ω χώριο οτοκία και γι' αυτό δεν υπάρχουν και κοινέ συστάσει, κυρίω ε, βάσει του άρθρου 8, γιατί υπάρχουν οι ίδιε αντιρρήσει που υπάρχουν στα πλαίσια των συζητήσεων που, γίνεται, που γίνονται υπό το άρθρο 11. Ευχαριστώ. Ίσως να πρέπει να το ξέρω αυτό, αλλά αυτή η περιοχή της ανάκτησης, αν ε, οριστεί άπαξ, ε, μπορεί να αλλάξει ή θα υπάρχει για πάντα τι σημαίνει για τις χώρες που πρέπει να τις ε, ορίσουν αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, αν γίνει κάποιο λάθος μια φορά, μετά τι γίνεται, καταδικάστηκαν για το υπόλοιπο της ζωής τους, οι στοδιειναικές. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σημεία θέλω να θίξω. Καταρχάς, στη Βόρεια Θάλασσα έγινε μία προσπάθεια το 2018 για την καλλιέργεια στριβιών σε μια περιοχή που ήταν κοντά σε ένα ελληνικό πάρκο και 90% των στριβιών τελικώς δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν. Ήταν μια παρενέργεια την οποία δεν είχαμε υπολογίσει. Ε, μπορείτε να μας πείτε ε, κάτι σχετικά με αυτό. Επίσης, ένα πράγμα το 2018. Σε μια άλλη περιοχή, 80.000 στρίδια είχαν καλλιεργηθεί έτσι ώστε να ανακτηθεί η δυνατότητα παραγωγής τους. Μόνο τέσσερα στρίδια, γόνοι καταγράφηκαν εκεί. Και επίσης, δεν ξέρω αν μπορείτε πιο εύκολα να μας απαντήσετε γραπτός, μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και ένα ερώτημα από ένα συνάδελφο που δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα, από μία συνάδελφο, συγγνώμη, ε, για τις ε, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Ήθελε η συνάδελφος να ρωτήσω εάν αυτές οι περιοχές διασπούν τις ε, ε θαλάσσιες περιοχές σε αφύσικες σε αφύσικα τμήματα και περι, περιπλέκει την ε, θαλάσσια ίσως χαρτογράφηση. Ε, η Κομισιόν ενεργώς ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν την προσέγγιση αυτή και θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται και με την αεραστεχνική αλία και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμπεριλαμβάνει και αυτή στον υπολογισμό των κοινωνικο-οικονομικών ωφελών. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε στα δύο ερωτήματα. Um, ναι, να απαντήσω στην ερώτηση του ε, κυρίου Γκλάντης για το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Είναι μια κοινή σύσταση ε, με την οποία συμφώνησαν τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει καμία για το άρθρο 8. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ποια είναι η πρακτική, αλλά η πρακτική με βάση το άρθρο 11 είναι ότι αυτές οι, κοινε, οι, προβλέπουν μια ε, ρήτρα αξιολόγηση. Άρα αυτά τα μέτρα δεν θα είναι για πάντα. Ε, προκειμένου κάποια στιγμή να γίνει μια αξιολόγηση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και αν είναι ε, τα κατάλληλα μέτρα. Υπάρχει λοιπόν μια ρήτρα αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κύριου Φαντάλενς για το αιωλικό πάρκο στην Βόρεια Θάλασσα, δεν γνωρίζω κάτι σχετικά. Ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει πρόβλημα με τις θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες όταν παίρνουμε μέτρα που αφορούν μόνο την αλληλεία αν λέμε απαγορεύουμε απλώς την αλεία, αλλά επιτρέπουμε τις εξορίξεις, ε, υπάρχει πρόβλημα. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση όταν καθιερώνουν τέτοιες ζώνες στα κράτη-μέλη. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να προστατεύσουμε, πώς θα το καταφέρουμε. Πρέπει να πάρουμε ε, μέτρα που αφορούν και την αλεία και άλλες ε, διαστάσεις στα πλαίσια των κοινών συστάσεων. Εμείς ε, αξιολογούμε τα μέτρα αλίας, γιατί δεν έχουμε την, ε, την αρμοδιότητα να αξιολογήσουμε τα αιωλικά πάρκα, αλλά είναι πολύ καλή ε, ερώτηση για το σχεδιασμό. Στη Βόρεια Θάλασσα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα, κυρίως με τα ε, αιωλικά πάρκα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένας καλός ε, θαλάσσιος σχεδιασμός. Σε ό,τι αφορά τη διάσπαση των θαλάσσιων ζωνών, ε, πώς μπορούν να καθοριστούν οι προστατευόμενες ζώνες. αυτό το θέμα τίθεται. Έχουμε έναν στόχο. Δεν είναι μόνο 10% προστατευόμενων ζώνων, ζωνών. Ε, πρόκειται για ένα δίκτυο ζωνών, δεν πρόκειται για ε, μεμονωμένες ζώνες. Πρέπει να ε, συνδέονται, πρέπει ο στόχος να είναι γενικός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέμορη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν κάποια ζώνη χρειάζεται ανάκτηση των ε, αποθεμάτων είναι αυτές που έχουν υποστεί ε, ηλεκτροπληξία από τους ε, Ολλανδούς. Αυτή η πρακτική έχει απαγορευτεί σε άλλες χώρες, στην ΣΥΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, το Καναδά και στην Βραζιλία. Και αν κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για το ε, ε, περιβάλλον, γιατί αφήνει τους Ολλανδούς να μοιράζουν τέτοιες άδειες και να ε, αγνοούν νομοθεσία και να προβάλλουν σε τέτοιες πρακτικές. Αντί να τηρούν τους, τα όρια που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ε, πρακτικές των ε, Ολλανδών κάνουν το θαλάσσιο βυθό να φαίνεται σαν έρημο και έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματα των ψαριών. Ε, οι ποσότητες γλώσσας και άλλων ψαριών έχουν μειωθεί δραματικά και οφείλονται σε αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί πώς τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες ε, συζητήσεις όταν γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ε, πρακτικών τους ε, για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το τι βγάζουμε από το νερό, αλλά και πώς επηρεάζουμε, τι ζημιά κάνουμε στο περιβάλλον μελέτες του Βρετανικού Οργανισμού ΣΥΦΑΣ έχουν αναδείξει αυτή την πρακτική ως μια πολύ επικίνδυνη πρακτική, η οποία πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μέμορη. Δυστυχώ θα πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Βαντέλε μετά το τέλο τη συζήτηση, γιατί αλλιώ θα αρχίσουν να βγαίνουν ατμοί από το κεφάλι του. Ε, γιατί τον εκνευρίσατε. Κύρια Οσάλεβαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας ε, την τελευταία παρέμβαση, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει ε, εντατική ανάλυση με τους ενδιαφερομένους για να μπορέσει να ε, γνωρίζει κάποια πράγματα για τον όλο τομέα της ε, αλίας. Κύριε Πρόεδρε, εσείς αναφέρατε το 3% των MPAs και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι υπάρχει ένα στόχος του 10%. Πάρα πολύ λίγη λοιπόν ε, συμμετοχή σε σχέση με τα MPAs. Θα πρέπει να υπάρχει εδώ κάποιο κίνητρο, αναρωτιέμαι. Ξέρουμε ότι είναι καλή για την υγεία των ωκεανών, ξέρουμε ότι όπως πολλοί είπανε ότι είναι καλά για τα οικοσυστήματα. Όπως είπε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει ένας διάδρομος αποτελεσματικών MPAs, ε, πραγματικά υπάρχει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την παραγωγικότητα για τα αλληλευτικά αποθέματα. Επομένως, ε, στο δικό μου το μυαλό τα MPAs είναι κάτι τα οποία θα πρέπει ε, ε, να προσπαθεί να έχει ένα κράτος μέλος και πραγματικά ε, ε υπάρχουν ερωτηματικά γιατί δεν υπάρχει τόσο, υπάρχει τόσο χαμηλή συμμετοχή. Τώρα, εάν τα MPAs τα οποία έχουν εφαρμοστεί υπόκειται αρνητικέ συνέπειες από διάφορες αλληλεκτικές δραστηριότητες ε, μπορούμε να τα αποκαλούμε MPAs. Στη Βόρεια Θάλασσα, στη, στο Ντόβερ, υπάρχει ένα MPA και συζητάτε και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ε, κάποια ε, εξαρτήματα αλληλευτικά βαθέων υδάτων ε, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η οδηγία είναι πάρα πολύ σαφής ε, και αυτό ουσιαστικά παραβιάζει το τι θα πρέπει να είναι MPA. Ε, προβλέπεται ότι οι δραστηριότητες στο Natura 2000 ε, επιτρέπονται ε, μόνο εάν αποδεικνύεται πέραν πάσης επιστημονικής αμφιβολίας ότι δεν θα έχουν αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του MPA. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η αναθεώρηση των κοινών συστάσεων που υποβλήθησαν από ε, τα κράτη-μέλη θα βασίζεται στις ε, πιο επιστημονικές ενδείξεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το MPA θα τηρεί το πρότυπο του άρθρου 6 της Οδηγίας για τους Φυσικούς Σκοτόπους και ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος για το ευνοϊκό περιβαλλοντικό καθεστώς ή το ε, ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Ευχαριστώ κυρία Σάπρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στα δύο μέσα διακυβέρνησης. Δεν ξέρω πώς γίνεται η οργάνωση στα άλλα κράτη-μέλη. Στη Γαλλία έχουμε, ανεξάρτητα από το Natura 2000, ε, τα θαλάσσια πάρκα. Και επίσης, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη, πρέπει να γίνει σχεδιασμός ε, των θαλάσσιων χώρων, ε, το είπαν και οι συνάδελφοι από την εμπειρία που διαθέτω, γιατί ήμουνα στον οργανισμό των ε, θαλάσσιων περιοχών και πέρασα και αυτό στο σχεδιασμό των θαλάσσιων χώρων, τα δύο βασικά στοιχεία είναι αυτών των μέσων διακυβέρνηση είναι ότι υπάρχει μια επιτροπή διαχείριση. Δηλαδή, ο καθορισμένος θαλάσσιος χώρος ε, είναι αντικείμενο συνδιαχείρισης με όλους τους συμμετέχοντες και οι περιοχές οι οποίες πρέπει να προστατεύονται καθορίζονται συλλογικά, ε, λαμβάνονται τα μέτρα κλπ. Και θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης μπορεί να αποτελεί και εγγύηση αφενός ε, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, ε, του καθορισμού των ζωνών που θα πρέπει ε, να προστατεύονται ή να ενισχύεται η προστασία τους και ακόμα και αυτά τα μέσα διακυβέρνησης, αυτά τα θαλάσσια πέαρκα ε, μπορούν να τα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια παρακολούθηση και να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται το θέμα. Η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι και για το σχεδιασμό είναι λίγο το ίδια πράγματα, είναι ότι αυτή τη στιγμή μια προστατευόμενη περιοχή έχει ένα ε, κοινό εργαλείο διαχείρισης ε, και έχουμε και τους ενδιαφερομένους, ε, οι επιστήμονες, οι κυβερνητικές οργανώσεις, ο οικονομικός κλάδος, αν λοιπόν είναι όλα επιμερισμένα, είναι κάτι που έχουν οικοδομήσει όλοι από κοινού και πιστεύω ότι έτσι τα πράγματα ε, τα διαχειριζόμαστε και πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Ε, τα θαλάσσια πάρκα και ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε στη Γαλλία θεωρείται ότι είναι ε, ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού. Τι γίνεται δηλαδή με τα θαλάσσια πάρκα και τον προγραμματισμό. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε che. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μέχρι το 2020 το στόχο να εγγυηθούμε το 20% των ε, παράκτιων περιοχών που είχε ε, καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα στοιχεία τα οποία μας ε, εντυπωσιάζουν είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου διαφάνεια για τις προστατευόμενες περιοχές στα κράτη-μέλη και υπάρχουν χρόνιες καθυστερήσεις ε, για την εισαγωγή των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων. Και να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά είναι τα κράτη-μέλη ή και ένα σύστημα που είναι οδηγία, επόμενη οδηγία και αλλάζουν οι αρμόδιες αρχές και οι βάσεις δεδομένων και τελικά είναι πολύ πολύπλοκο και πρέπει κάπως να το απλουστεύσουμε. Μετά, λαμβάνω και κάποιες επιστολές από κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θίγουν κάποιες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ε, η ε, βιομηχανική αλληλεία μετράτες γίνεται κατά 1,2% περισσότερο από ό,τι τις, ε, στις μη προστατευόμενες περιοχές. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι παράλογο το να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διότι, ε, αλληλιακή, διότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ε, κανονικά θα έπρεπε να είναι ένας χώρος ο οποίος ε, αποτελεί ε, ένα όνειρο και θα πρέπει να το προστατεύουμε. Τι γίνεται λοιπόν και επίσης τι γίνεται με τις τοπικές αρχές και τις προστατευόμενες περιοχές. Και επίσης κάτι τελευταίο, η ΜΚΟ και πάλι ε, μας ρωτούν αν σκοπεύετε να λάβετε υπόψη την απαγόρευση καταστροφικών πρακτικών αλίας εντός των ίδιων των προστατευόμενων περιοχών. Uh, I just um, Δύο ακόμα μιλητέ. Έχω τον κύριο Μιγιάν και τον κύριο Βαντάλεν. Αν δεν σα πειράζει, να ακούσουμε όλε τι ερωτήσει και μετά να ε, απαντήσετε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Αναφερθήκατε σε μία έκθεση του ΣΥΦΑΣ. Από ό,τι φαίνεται οι εκθέσεις τους δημοσιεύτηκαν προσφάτως ε, είδα λίγο την ε, σύνοψη η οποία ε, δεν είναι και πολύ επιστημονική. Λέει από τη μια έχουμε αυτό και από την άλλη το άλλο και θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα. Ο κύριος Βαντάλεν. Προφανώς και ήθελα το λόγο για να απαντήσω στα όσα είπατε. Από τη μια έχουμε το Brexit και από την άλλη έχουμε την Αλία και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά ψεύδι που πλανώνται στον αέρα για τα δύο αυτά πράγματα. Οι, οι υπέρμαχοι του Brexit ε, μας ταΐζουν εδώ τα ψεύδι τους καθημερινά, αλλά η κυρία αυτή μας ανέφερε διάφορα ψεύδι εδώ σήμερα το απόγευμα. Άνθρωποι που έχουν βρεθεί εδώ στην Επιτροπή θα έχουν... Ε, υπόψη τους ότι ήρθε ο πρόεδρος τη Επιτροπής ISIS και μίλησε για επιστημονικέ γνωμοδοτήσεις και είπε σαφέστατε επανειλημμένος ότι επί τη βάση μελετών ότι υπάρχουν ε, ε, πλο, ε, ωφέλη σε αυτή τη μορφή αλληλείας μέσω ε, ηλεκτροπληξίας και ότι είναι πολύ πιο ευνοϊκή σε σχέση με την παραδοσιακή τράτα. Υπάρχουν πολλά ψεύδη τα οποία κυκλοφορούν από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους και λένε για παράδειγμα ότι ε, το 1,5% ε, των ε, οστών του γάδου καταστρέφονται από την αλία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η καταστροφή είναι από την συνήθι μορφή αλίας με τράτα και όχι με την ε, μορφή αλίας με ηλεκτροδότηση τα επιστημονικά γεγονότα αποδεικνύουν εντελώ το αντίθετο από αυτά τα οποία ισχυρίστηκε η συνάδελφο. Εγώ είμαι υπέρμαχο λοιπόν τη επιστημονική άποψη, δεν είμαι υπέρμαχο του Brexit και θα ήθελα να αποσύρει τα σχόλιά του η συνάδελφο. Όπω σα είπα, κάποια μέλη που ήταν εδώ στην προηγούμενη θητεία θα τα έχουν ξανακούσει αυτά τα επιχειρήματα. Εγώ έριξα μια σύντομη ματιά σε αυτή τη μελέτη και λέει αφενός υπάρχει αυτό και αφετέρου υπάρχει το άλλο. Κάτι το οποίο ένας ε, θεωρεί ψέμα, ο άλλος μπορεί να το θεωρεί όχι. Ε, Κυρία Μέμορη, όχι αυτή τη φορά. Ε, θα μείνουμε στις προστατευόμενες περιοχές. Ε, ο κύριος Μηγερμόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι περιοχές θαλάσσιας προστασίας είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση όχι μόνο των θαλασσών, αλλά και της βιοπικιλότητας και πιστεύω ότι αυξάνεται στην Ευρώπη και έχω ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σύμφωνα με τις πληροφορίε που έχω, το 2001 στην Ισπανία είχαμε περίπου το 1% των ακτών που είχαν αυτό το χαρακτήρα των ε, προστατευόμενων ζωνών. Και πλέον είμαστε ήδη στο 10%. Τουλάχιστον στη χώρα μου λοιπόν υπήρχε μεγάλη πρόοδο ε, για να, ανακηρυχθούν κάποιε περιοχέ, προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχέ. Ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλε φιλοδοξίε διεθνώ και ε, ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες προωθούν πάρα πολύ αυτή την ε, σύνοδο βιοπικιλότητας και υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες, αλλά τουλάχιστον για το 10% στη χώρα μου επετεύχθη. Ο στόχος για το 2020 είναι ε, λοιπόν ε, ήδη αυτό που περιμέναμε. Commission, can we, can we turn to you to respond? Commission, να απαντήσετε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο. Καταρχά για τι περιοχέ ε, ε, ε, ανάκτηση, πόσε έχουν δηλωθεί, καμία, μηδέν. Για το άρθρο 11 πάλι ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Απ' την άλλη, όπω είπε και ο κύριο Μιγιανμόν, πολλές περιοχές θεωρούνται ε, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και ελάχιστε έχουν και σχέδιο διαχείριση οι περιοχές αυτές έχουν ε, δηλωθεί ως τέτοιες, όχι για να προστατεύσουν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, ή όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να δώσουν ε, ε, πλεονέκτηματα στην αλλιευτική βιομηχανία για να υπάρχουν χώροι οτοκίας ηχθείων. Νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε λίγο περισσότερο τα κρατημέλη να βάλουν λίγο ζουμί σε όλα αυτά τα θεωρητικά. Εντάξει, καλοί είναι οι χάρτες, αλλά αν δεν έχουμε διαχείριση και πρακτικά αποτελέσματα, δεν οφειλούν σε τίποτα. Οπότε μήπως πρέπει να μα πείτε πώς μπορούμε εμείς να πιέσουμε εσάς να κάνετε περισσότερα. Εγώ θα έλεγα να πιέσετε τα κράτη-μέλη περισσότερο. Ναι, εντάξει, αλλά εσείς έχετε τη νομική δύναμη να το κάνετε αυτό. Ποιος καλύτερος από εσά. Ε, θα διαφωνήσω. Ε, δεν έχουμε τόσες μεγάλες ε, δυνατότητες. Βεβαίως η Κομισιόν ακούει τα κρατημέλη, αναλαμβάνει το ρόλο της διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας, αλλά τι μπορεί να γίνει παραπάνω, ε, δεν τα έχουμε παρατήσει. Εντάξει, δεν τα παρατάει η Κομισιόν. με κάθε εργαλείο που έχουμε προσπαθούμε να πιέζουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι παραπάνω για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να διαχειριστούμε καλύτερα τις περιοχές αυτές, βεβαίως μέσα στα εργαλεία που έχει να μας δώσει η κοινή ελευτική πολιτική. Να πάω πίσω τώρα στα ερωτήματα που πήραμε από την κυρία Οσάλιβαν για τις επιστημονικές, ε, τα επιστημονικά στοιχεία και τις κοινέ συστάσεις για το πώς θα αξιολογηθούν στα πλαίσια της ε, επιστημονικής αξιολόγηση. Είναι ε, τρέχουσα, στάνταρ συγγνώμη διαδικασία, ίσως να μην το είπα. Ε, όποτε λαμβάνουμε μια τέτοια μεικτή κοινή σύσταση από τα κρατημέλη, πάντα αξιολογείται από την Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή για την Αλληλεία. Και αυτή η Επιτροπή πρέπει να μας πει κατά πόσο αυτή η κοινή σύσταση πληρεί μπορεί να επιτύχει το στόχο και αν μπορεί να συμβάλλει για την επίτευξη των στόχων της, νομοθε... της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αν δηλαδή είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην πρώτη μου παρέμβαση. Σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν μπορεί να επιτύχει από μόνη τη η σύσταση την ε, ναι, περιβαλλοντική νομοθεσία. Πρέπει όμω να μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Και αυτό κάνει η STCF. Αυτό αξιολογεί. Αν είναι βήμα προ τα εμπρό. Τώρα, για τα όσα είπε η κυρία Σαμπό για την ε, συμμετοχή των ε, μπλεκόμενων φορέων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και στη δική μας την επαφή με τα κράτη-μέλη σε όλη αυτή τη διαδικασία πάντα τα ενθαρρύνουμε να, να βάζουν από την αρχή της διαδικασίας στο παιχνίδι του εμπλεκόμενους φορείς. Αν, αν ληφθούν μέτρα χωρίς τη στήριξή τους, χωρίς ε, τις βασικές ε, κοινωνικές ομάδες θα είναι αποτυχία. Γι' αυτό θα τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν. Αλλά βεβαίως πάλι οι περιφερειακές ομάδες είναι αυτές που πρέπει να δουν πώς θα την προσεγγίσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν με την εμπλοκή των, των εμπλεκόμενων φορέων, όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να πάνε στο συμβουλευτικό ε, σώμα. Οπότε και εκεί μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση για του ε, εμπλεκόμενου φορεί. Και εκεί δηλαδή μπορούν να μιλήσουν για τη σύσταση αυτή οι εμπλεκόμενοι φορέ. Αλλά βεβαίω καλύτερο είναι να έχουν συμμετάσχει από την αρχή. Και ξέρουμε ότι στι περισσότερε περιπτώσει υπάρχει συμμετοχή του από την αρχή. Πρέπει να πω ότι, η... μάλλον δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Κάθε περιφέρεια έχει τα εργαλεία να δει τις ιδιαιτερότητες ε, που την ε, διέπουν. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια λύση για όλους. Καλό θα ήταν η κάθε περιοχή να ορίσει τι είναι καλύτερο για αυτή. Και για τα όσα είπε η κυρία Νταμάτο, να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλερή Λενέ για να απαντήσει. Ε, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο πράγματι, η κυρία Σαμπό έχει ε, δίκιο. Υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα, αλλά ελήφθησαν και κάποια μέτρα από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της εφαρμογής του ε, κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα για τη Μεσόγειο. Ε, καθιέρωσαν λοιπόν ζώνες προστασίας ε, που εντάχθηκαν στα εθνικά σχέδια δράσης. Εφαρμόστηκαν κάποια σχέδια που προβλέπουν κάποιες ζώνες προστασίας στα ε, εθνικά ύδατα. Ε, η Ισπανία είναι ένα παράδειγμα όπου η καθιέρωση αυτών των ζωνών έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για την προστασία των γόνων και των ευαίσθητων περιοχών. Πολύ θετικά τα παραδείγματα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Η Κομισιόν θα κάνει μία χαρτογράφηση και θα την δημοσιεύσει του χρόνου για την Μεσόγειο, προκειμένου να αναδειχτούν τα μέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό ε, επίπεδο για την προστασία των ε, ευάλωτων ενδιατημάτων και των γόνων. Αυτό θα προσφέρει μια διαφάνεια, θα φανούν οι προσπάθειες που έχουν ε, καταβληθεί. Σε επίπεδο της GFCM αποφασίστηκε ότι η Γραμματεία θα προβεί σε μια αξιολόγηση των μετρών, ε, μέτρων ε, στις ζώνες ε, προστασίας προκειμένου να δούμε αν είναι αποτελεσματικά ή όχι. Α, τι μέτρα θα μπορούν να ληφθούν στο μέτρο, να εναρμοζηστούν τα μέτρα στις ζώνες προστασίας και να ενισχυθούν. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα πιλωτικό πρόγραμμα με τη χρήση ενός δορυφορικού προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να προστατευτούν οι δραστηριότητες σε αυτές τις ζώνες προστασίας. Στη Μεσόγειο λοιπόν ε, υπάρχει μία δραστηριο, ε, δραστηριοποίηση και όσο πιο διαφανής είμαστε, τόσο περισσότερο θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και διάφοροι φορείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Σαμπό. Ε, χρειαζόμαστε μία συμμετοχική προσέγγιση ε, δηλαδή χρειαζόμαστε τη συμμετοχή και των αρχών και των επιστημόνων και των αλλιέων και όλων των φορέων. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ε, να επαναλάβω το παράδειγμα που σας, έδω, σας έδωσα με τη συμμετοχή τριών ε, παραγόντων και έτσι επιτύχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έτσι επιτύχαμε την εφαρμογή των μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που ε, θα συνεχίζουν να ασκούν πίεση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο ε, η Συμφωνία ε, Σύμπραξης με την Γκάμπια. Το Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο να υπογράψει αυτήν την συμφωνία, αλλά λάβαμε την ε, απόφαση εσύ προς έγκριση τον ε, Αυγούστο. Η κυρία με ορίστηκε η συγκήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, ε, πρόκειται για τα συμπεράσματα για την σύναψη συμφωνία σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γκάμπια. Η Γκάμπια είναι μία από τις μικρότερες χώρες ε, της Αφρικανικής Υπήρου ε, στις όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού και είναι μία από τις πιο πλούσιες αλληλευτικές ζώνες στον κόσμο. θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την, τον αλληλευτικό κλάδο για την Κάμπια, όμως αυτός ο κλάδος συμμετέχει πολύ λίγο στην ανάπτυξη της χώρας και αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή διαχείριση των αλληλευτικών πόρων, την ανεπαρκή επιστημονική έρευνα και τα υψηλά επίπεδα παράνομης λαθρέας και ε, άναρχης αλίας. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ε, υποτίμηση των στοιχείων της αλίας στην ε, Γκάμπια. Γι' αυτό ήταν απαραίτητη η σύναψη μια συμφωνία σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γκάμπια, προκειμένου η ε, χώρα να μπορέσει να, ανακτησει βημα ε, βήμα-βήμα τον έλεγχο των αλευτικών πόρων της. Πρόκειται για μια νέα συμφωνία που αντικαθιστά την προηγούμενη, ε, η οποία ε, τέθηκε σε ισχύ το 1987, η οποία έχει λήξει όμως. Ε, το νέο πρωτόκολλο καλύπτει μια εξιετή περίοδο και λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, τις εξορετικές ε, διαστάσεις και τη δράση των κοινοτικών ε, των ευρωπαϊκών σκαφών στα ύδατα της Γκάμπια, προωθώντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη αλληλευτική πολιτική και διαχείριση των αλληλευτικών πόρων ε, στα ύδατα των δύο μερών. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία ε, δίνει τη δυνατότητα ε, στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να αλλιεύουν περίπου 300.000 τόνους τόνο στα ύδατα της Γκάμπια και 400.000 τόνους μπακαλιάρου. Η προβλέπει ενίσχυση της διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων και του αλληλευτικού κλάδου στην ε, Γκάμπια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πληρώνει 17 ευρώ ανατόνο τόνο τόνου στην Γκάμπια. Ε, εγώ θα ήθελα να απευθύνω ερώτημα στην Γενική Διεύθυνση, απεύθυνα ερώτημα στην Γενική Διεύθυνση ε, Θαλάσσιας Πολιτικής ε, για το χαμηλό ε, ποσό αυτής της τιμής. Η απάντηση ήταν δόθηκαν κάποιες απαντήσεις ε, ελήφθησαν υπόψη δραστηριότητες παράνομης, λαφρέας και άναρχης αλίας. Επίσης η Γκάμπια δεσμεύτηκε να ε, συμμετάσχει στον, στις δράσεις του ICCAT είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία και το πρωτόκολλο εφαρμογής και για την ε, Γκάμπια και για τα... το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται στα ύδατα της ε, Γκάμπια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία για τα αποθέματα στην περιοχή και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά σκάπη δεν θα συμβάλλουν στην ε, υπεραλίευση. Σίγουρα θα ε, δαπανηθούν τα κονδύλια έτσι όπως ε, προβλέπετε και πώς θα αποφευθεί η αλίευση γόνων. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να επαναλάβετε την τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Κυρία Βαντέλα. Ποια είναι τα να ξαναρχίσω. Ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία για τα αποθέματα στην περιοχή και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά σκάφη δεν θα συμβάλλουν στην υπεραλίευση. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την αλίευση του τόνου, πώς θα αποτρέψουν την αλίευση γόνων και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια θα δαπανηθούν σύμφωνα με τους ε, καθορισμένους στόχους. Όλα τα στοιχεία, τα επιστημονικά στοιχεία μας δόθηκαν από την ε, Γενική Διεύθυνση Αλίας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει έλεγχο κάθε ε, σκάφους και τις σχετικές διαδικασίες οποιοδήποτε ψάρι θα λιεύεται στα ύδατα της ε, Γκάμπιας, ε, της Γκάμπια. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι ήδη δραστηριοποιούνται ευρωπαϊκά σκάφη στα ύδατα της Γκάμπια και υπάγονται στους προβλεπόμενους ελέγχους. Κυρία Βαντέλα. Η ομάδα μας όρισε την κυρία ε, Σαγιάννερ Μάριμ για ως ε, σκιώδη εισηγήτρια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την συμφωνία. Το είπε ξεκάθαρα η εισηγήτρια και θα ήθελα να το επαναλάβω σε ό,τι μας αφορά την Κάμπια ε, είναι πλούσια τα ε, ηχθιαποθέματα, είναι υψηλή η βιοπικιλότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να την προστατεύσουμε και Φυσικά πρέπει να ε, επιμείνουμε στη σημασία της καταπολέμησης της παράνομης λαθρέας και ε, άναρχης ε, αλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να υποστηρίξει την Κάμπια στην προσπάθεια της διατήρησης της βιοπικιλότητας. Στο όνομα λοιπόν της Κιόδους εισηγήτριας θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για την παρουσίαση της σύνοψης της έκθεσης, ε, η οποία είναι πολύ ικανοποιητική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γκάμπια είναι ένα καινούριο ε, μέλος των, στην όλη προσπάθεια για χείριση της αλίας. Ε, πρόσφατα εντάξαμε λοιπόν την Κάμπια στην ε, όλη προσπάθεια διαχείρισης της ε, αλληλευτικής πολιτικής. Ε, η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, στη διαφάνεια, λαμβάνουμε υπόψη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η κεντρική στόχη μας και αντικατοπτρίζονται πλήρως στην ε, συμφωνία και στο πρωτόκολλο εφαρμογής της που υπεγράφησαν με την Γκάμπια. Για να επανέλθω στα ερωτήματα που έθεσαν οι διάφοροι συνάδελφοι, η οικονομική διάσταση δεν ε, πρέπει να λάβουμε, υπολογίσουμε 70 ευρώ το τόνο, αλλά 120 ευρώ ανατόνους. Οι ε, πλη, ε, πλειοκτήτες ε, θα ε, συμμετέχουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει 50 ευρώ ανατόνο. 120 ευρώ λοιπόν ανατόνο θα πηγαίνουν στην Κάμπια. Άρα και ε, επίσης ε, οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο των αλλιευμάτων, το ε, κομμάτι που αναλογεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πηγαίνει πάντα στην, συστηματικά στην γκάμπια. Και αν αξιολογήσουμε αυτά τα, συγκρίνουμε αυτά τα 120 ευρώ τόνο με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές, ε, ξέρουμε ότι το ποσό συνάδει με τα, ε, τις υπόλοιπες συμφωνίες που έχουμε συνάψει σε αυτή την περιοχή και με τις επενδύσεις ε, που πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τον, τη διαχείριση των αποθεμάτων του τόνου. Πρέπει επίσης να διακρίνουμε από τη μία τα αποθέματα των θηνοειδών, η κατάσταση των αποθεμάτων είναι καλή, ε, αξιολογούνται σε περιφερειακό επίπεδο από τον ICCAT. Το Νοέμβριο ε, θα γίνει η ολομέλεια αυτής της οργάνωσης. Έχουν ληφθεί μέτρα διαχείρισης που ίσως ε, ενισχυθούν και αυτά τα μέτρα διαχείρισης θα ε, αφορούν και τους ευρωπαϊκούς στόλους που θα δραστηριοποιηθούν στα ύδατα της Γκάμπια και των άλλων χωρών της περιοχής. Σε ό,τι αφορά το ε, μπακαλιάρο της ε, Σενεγάλης, είναι περιορισμένες οι, περιορισμένος ο αριθμός των σκαφών, δύο συγκεκριμένα θα υπάρχει ένας ε, παρατηρητής, ε, ε, είναι μια δοκιμαστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα αποθέματα του μπακαλιάρου της Σενεγάλης. Τέθηκε το ερώτημα των αλληλευτικών πρακτικών και των επιπτώσεων στους γόνους. Αν κοιτάξουμε τα σκάφη αλίας τόνου ε, τηρούν τις προδιαγραφές ε, για ε, τα σχετικά σκάφη. Θα έχουμε 20... Θα έχουμε συγκεκριμένο αριθμό σκαφών αλίας θηνοειδών που θα ε, τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ό,τι αφορά τις ε, τη διαχείριση των αποθεμάτων και την προστασία των ε, γόνων. Και ε, ο ΙΚΑΤ θα δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Ελπίζω να έδωσα από την πλευρά μου απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους υποστηρίζουν την συμφωνία. Έχουμε ήδη μια συμφωνία με την Σενεγάλη. Ε, ε, διαπραγματευτήκαμε μια, ένα νέο πρωτόκολλο και είναι σημαντικό να υπάρχουν ε, τέτοιες συμφωνίες ταυτόχρονα και στη Σεναγάλη και στην Γκάμπια, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι δεν θα υπάρχει υπεραλίευση και δεν θα αλλιεύονται γόνοι. Αυτό που ε, εφαρμόζουμε είναι μέτρα ελέγχου. Η δέσμευση είναι των κρατών ε, μελών να τηρούν τους ε, κανόνες που προβλέπονται από την νομοθεσία της Γκάμπια, τη Συμφωνία Σύμπρεξης και σε περιφερειακό επίπεδο. Αν υπάρχει περιέλευση των θηνοειδών, αυτό πρέπει να αξιολογηθεί από τον ICCAT και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συζητηθούν τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά τον μπακαλιάρο της Εναγάλης, είναι ε, πολύ συγκεκριμένα και ελεγχόμενα τα πλαίσια και μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για μια ενδεχόμενη υπερελίευση του συγκεκριμένου είδους στα πλαίσια αυτή της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα, ήθελ, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών ε, ε, η Παρασκευή, 12 η ώρα. Αύριο το πρωί θα έχουμε μια σύντομη συνάντηση. Σήμερα το βράδυ ε, μπορείτε να έρθετε ε, στη συνάντηση που θα έχουμε με τις ε, ΜΚΟ σχετικά με το θέμα της παράνομης λαθρείας και άναρχης αλίας. Θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ. Στις 6.30 ξεκινάει η συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.